Good morning, ladies and gentlemen. May I ask... Καλημέρα σας, παρακαλώ να καθίσετε. We have a busy program in the morning. Κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολλά πράγματα για συζήτηση στην πρωινή συνεδρίαση και γι' αυτό θα ήθελα να μην καθυστερήσουμε άλλο. Αρχίζουμε λοιπόν. Σύμφωνα με την υπηρεσία διάταξη θα ξεκινήσουμε με την αποστολή το Σεπτέμβριο στο Κλους Ναπόκα και στη Σόφια τον Οκτώβριο. Υπάρχει κάποιος από τους συναδέλφους που πήραν μέρος στο κλούς να πόκα να πάρει το λόγο. Ο κύριος Βανίστελ Ρόι. Σύντομος παρακαλώ. Κοιτάξτε, μας άνοιξε πολύ στα μάτια αυτό που κάναμε. Ήμασταν καλά προετοιμασμένοι, είχαμε συναντήσεις και με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είχαμε στοιχεία, συναντηθήκαμε με υπουργούς και αυτά όλα μας έδειξαν ότι αρκετά πράγματα έχουν αλλάξει κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και ιδιαίτερα στην περιοχή του Κλούς την τη βόρειο-δυτική περιοχή της ε, Ρουμανίας. Αυτό το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι ότι η Ρουμανία μπορεί να, θα έλεγα, να ακολουθήσει μία πολιτική από το κέντρο της ε, ε, πολιτικής εξουσίας αλλά πρέπει να διαχειριστεί τις περιφέρειες της χώρας με τρόπο τέτοιο που να μην τους δημιουργεί ε, εμπόδια, να μην αποτελεί τροχοπέδι για την εξέλιξή τους και για τις ε, αποφάσεις των τοπικών περιφερειακών αρχών. Και εδώ ίσως ε, υπάρχει το πολωνικό παράδειγμα. Το πολωνικό παράδειγμα μας δείχνει ότι έχουν προχωρήσει σε τέτοιου είδους θέματα στο επίπεδο NET 2 και συζητούν θέματα όπως ας πούμε ε, περιφερειακές αρχές οι οποίες συνεργάζονται μεν μεταξύ τους αλλά όταν είναι μπροστά στην κεντρική εξουσία, στην ουσία είναι αδύναμες οι περιφερειακές αυτές μορφές εξουσίας. Και αυτό δημιουργεί ένα θέμα. Βλέπουμε λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο προχωρά η χώρα αυτή σε, με ένα επίπεδο δια, διακανονιστικό, ρυθμιστικό, αρκετά περίπλοκο. Το δεύτερο που πρέπει να πω είναι ότι η πόλη του Κλούς και οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, των πανεπιστημίων, του επιχειρηματικού κόσμου, της κοινωνίας των πολιτών έχουν σαν στόχο να δώσουν μια νέα όθηση σε νέες μορφές ανάπτυξης σε αυτό το τμήμα της χώρας. Εμείς επισκεφθήκαμε νέες επιχειρήσεις που πήγανε στο κλούς, η Μπός ας πούμε έχει ένα τμήμα της έρευνάς της εκεί για τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς για δίκυκλα χωρίς οδηγούς, δεν κατάλαβα και πάρα πολλά πράγματα και για ποδήλατα, δεν ξέρω, συνδεδεμένα ποδήλατα. Ελπίζω να έχουν οδηγό τα ποδήλατα, λέει ο κ. Νίστελοϊ. Και αυτό μας έδειξε ότι υπάρχει ζήτηση εκεί, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός φοιτητών σαν παράδειγμα που συγκεντρώνονται στην πόλη του Κλούζ. Και οι καταστάσεις αυτές είναι χρήσιμες για τους νέους της Ρωμανίας και η πόλη του Κλούς θέλει να δημιουργήσει και νέα κάμπους, θέλει να εντατικοποιήσει τις ερευνητικές αυτές δραστηριότητες γύρω από την πόλη και μπορέσαμε να δούμε πως οι τοπικές αρχές, οι τοπικές πρωτοβουλίες, οι περιφερειακές πρωτοβουλίες μπορούν να λειτουργήσουν στα πλαίσια της λεγόμενης νέας οικονομίας. Αυτό το είδαμε και στις μεταφορές, στις υποδομές τις συγκοινωνιακές που χρηματοδοτήθηκαν φυσικά από τα ταμεία συνοχής και νομίζω ότι καταλάβαμε πολλά. Δεν διάβασα την τελική έκθεση ακόμα. Νομίζω πάντως ότι πρέπει να ευχαριστήσω αυτούς που το οργάνωσαν. Εντάξτε, μόλις ήρθα έτσι κι αλλιώς. Έπρεπε στις 8.30 το πρωί να ψηφίζω στην ΕΚΟΝ, οπότε τώρα μόλις μπήκα, μη με παρεξηγείτε, πάντω νομίζω ότι η δουλειά που έγινε στην αποστολή αυτή ήταν πολύ θετική. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα κυρία Κρέλ να κάνω μια παρατήρηση. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η αποστολή γιατί είδαμε μια περιφέρεια ουσιαστικά, όχι μόνο μια πόλη. Ήρθαμε σε επαφή με τους δημοτικούς συμβούλους ε, που έχουν πολλά να κάνουν. Ε, συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε ο Λάμπερτ Φανίστελ Ρόι, αλλά αποκόμισα και μια συγκεκριμένη εμπειρία που έτσι, με έχει κάπως προβληματίσει. Εμείς ε, ε, συνεργαζόμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαστε προσανατολισμένοι στα αντικειμενικά ζητήματα και αυτό τις περισσότερες φορές ε, ανεξάρτητα από την πολιτική μας ομάδα, τη χώρα μας κτλ. Αλλά στην Κλούζ, στην περιφέρεια της Κλούζ, η κυβέρνηση με τους υπουργούς όταν συναντάται με τους δημοτικούς συμβούλους και παλιά ήταν στην κυβέρνηση αυτή και ο ένας κατηγορεί τον άλλον ότι δεν λειτουργεί εφαρμογή λόγω των λαθών των προηγούμενων ή των νυν κτλ. Αυτό δεν βοηθάει καθόλου. Φυσικά ε, δεν είμαστε εμεί σε θέση να δίνουμε συμβουλές, αλλά τουλάχιστον καλό θα ήταν να υπάρχει έστω πιο καλή επικοινωνία, γιατί αυτό μπορεί να απελευθερώσει το δυναμικό της περιφέρειας. Στη Ρουμανία πραγματικά υπάρχει κεντρική διοίκηση, και κεντρική διαχείριση. Αυτό μας λυπεί εμά, αλλά είναι δική του απόφαση. Τουλάχιστον αν υπήρχε καλύτερη συνεργασία, ε, θα ήταν καλύτερα. Δεν ξέρω αν μπορούσαμε να το συμπεριλάβουμε κάπου στην έκθεση αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Βαν Ευχαριστώ. Ένα σύντομο σχόλιο να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στη Γραμματεία και στον κύριο Ντάνιελ Μπούντα, στην, στο Λορέντσιο, στην Κλάρα, στους ε, βοηθούς και στον Μπόγκταν που ήταν ο σύμβουλος πολιτικής μας, ο Ρουμάνος. Πραγματικά μας βοήθησαν να κάνουμε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα, το οποίο μου άνοιξε τα μάτια αντιλήφθηκα πως μια πόλη όπως η Κλουτζό μπορεί να αναπτυχθεί πραγματικά χάρη στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Κρίμα όμως ήταν ότι η κυρία Τζουφρίντα, η συγγήτρια της έκθεσης της Ρέτζη, δεν ήταν εκεί. Διότι εκεί είδαμε επί τόπου πόσο αναγκαίες είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα σωστό σύστημα διακυβέρνησης, και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα υγιές επενδυτικό κλίμα. Είδαμε ήδη την παρατήρηση του Lamberts, της Lamberts για αποκέντρωση, να λαμβάνονται αποφάσεις πιο κοντά στους πολίτες και εδώ βλέπουμε τα ωφέλη ενός κεντρικού συστήματος που σε ε, κάποιες ε, ε, περιπτώσεις δεν γνωρίζει τι κάνει, δεν θέλει να μεταρρυθμιστεί και που δημιουργεί προβλήματα στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και στις επενδύσεις. Για μένα, για άλλη μια φορά πρέπει να πω ότι αυτό η επίσκεψη μου άνοιξε τα μάτια. Πρέπει να δούμε τι συνέχεια θα δώσουμε ε, στις παρατηρήσεις, ε, στα διδάγματα που αποκομίσαμε αυτό το ταξίδι. Το θέμα δεν είναι να κάνουμε ένα ταξίδι κάθε δύο χρόνια σε κάποιες περιοχές για να παρακολουθούμε θα πρέπει να αποκομίζουμε και διδάγματα από τέτοια ταξίδια, να τα αποτυπώνουμε σε εκθέσεις. Οπότε υπολογίζω στην κυρία Κέλ ε, από τους σοσιαλιστές να συμπεριλάβει και, στη, σε μια εκθέση πληροφορίες για τις περιοχές που έχουν ε, μείνει ε, πίσω. Πιστεύω ότι ήταν μια πολύ επιτυχής αποστολή. Ευχαριστούμε κυρία Φάρα. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα και εγώ Συμφωνώ στα περισσότερα από όσα είπαν οι προλαλήσαντε συνάδελφοι, δύο μα είπε η κυρία Κρέλ. Επίσης και εγώ είδα κάτι ε, που δεν έχει αναφερθεί ακόμη. Πόσο μεγάλο δηλαδή είναι το χάσμα μεταξύ των προγραμμάτων και των στόχων της Ευρώπης 2020, δηλαδή των πολιτικών στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και υποτίθεται ότι αυτούς τους στόχους πρέπει να προωθούν και συνδέονται με αυτούς τους στόχους ε, τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται. Παραδείγματος χάρη, οδικές αρτηρίες, αυτοκινητόδρομοι που πραγματικά ε, παίρνουν πολύ μεγάλες επιδοτήσεις σε αντίθεση με τους αεροδρόμους και το συνδρομικό δίκτυο υπολείπεται τα μάλλα. Αυτό είναι κρίμα. Οι στόχοι 2020 είναι πολύ σημαντικοί και θα έπρεπε επιτόπου στο πρόγραμμα να τα αντικατοπτρίζεται αυτό. Ε, είδαμε επίσης ε, τα σχέδια για το προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού από το 7 στο ε, δεν ήταν και τόσο μεγάλη η πρόοδος εκεί και είδαμε και τις διοικητικές δομές ε, σε ό,τι ε, αφορά τη διοίκηση. Συμφωνώ με τους Σας Ευχαριστώ πρόεδρος κύριε Μπούντα. Πάρα πολύ σύντομα αν έχετε την καλωσή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που προετοίμασαν αυτή την αποστολή για την περιοχή του Κλούτζ ήταν πολύ σημαντική η παρουσία αυτής της αποστολής διότι ανταλλάξαμε εμπειρίε από τα όσα είπαμε εκεί πέρα. Ρίξαμε ένα νέο φως ε, στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την ανάπτυξη των περιφερειών. Γενικά ευχαριστώ όλους και πάλι που ήρθαν μαζί μα στο Κλούζ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για όλα αυτά τα σχόλια. Είναι πολύ σημαντικό που έχουμε συμπεράσματα από τις αποστολές μας αυτές. Η δεύτερη αντιπροσωπεία πήγε στην Σόφια στα τέλη Οκτωβρίου. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να μας ε, περιγράψει ε, τι, είδαν, τι είδε εκεί, κυρία Κρέλ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω θέρμα, κυρία Πρόεδρε που οργανώσατε αυτήν την επίσκεψη στη Σόφια. Για μένα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να δω τα διαφορετικά προγράμματα και των δύο περιόδων προγραμματισμού. Μπορέσαμε να επισκεφθούμε προγράμματα και από τις δύο περιόδους. Και επίσης ακούσαμε και ήταν ενδιαφέρον και για την προπαρασκευή της Βουλγαρικής Προεδρίας. Χθες στην Επιτροπή μας ακούσαμε για μια ακόμη φορά τα σχετικά ε, και πιστεύω ότι η βουλγαρική κυβέρνηση πράγματι ε, δίνει ιδιαίτερη σημασία ε, στην πολιτική συνοχή. Σε αυτό πιστεύουμε θα κάνει και στη διάρκεια της Προεδρίας της και πραγματικά πιστεύω σε πολλά σημεία θα έχουμε ένα πολύ ισχυρό εταίρο για να σημειώσουμε πρόοδο και να προετοιμάσουμε τη μελλοντική πολιτική συνοχή. Κάτι άλλο ενδιαφέρον που θέλω να αναφέρω ότι στην Σόφια την πρωτεύουσα αλλά και αλλού ε, στη Βουλγαρία. Υπάρχει πραγματικά ε, στο υπέδαφος ε, πλούτος πολιτισμικός και για την ε, ε, υλοποίηση κάποιων έργων, οδικών και λοιπόν πάντοτε πρέπει να γνωμοδοτήσει πρώτα η αρχαιολογική υπηρεσία και αυτό το είδα πάρα πολύ, έτσι, το θεώρησα πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί πρέπει να έχουμε υπόψη και την αρχαιολογία, την διατήρηση των πολιτιστικών μνημείων. Υπάρχει και ένα ποσό των 10 εκατομμυρίων που διατίθεται και ήταν πολύ ενδιαφέρον να δω ε, και τι γίνεται ε, με, τον πολιτισμό και τα σχετικά με τον κανονισμό Omnibus. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά που ε, οργανώσατε την επισκέψη αυτή. Πάρα πολύ καλή οργάνωση. Κρύο έκανε βέβαια, αλλά τέλος πάντων. <laughs> Αυτά είχαν από Πολύ καλή εμπειρία. Ευχαριστούμε πολύ ο κ. Βαν Μίλτεμπουργκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Κέρ στα όσα είπε. Να ευχαριστήσω επίσης ε, τη γραμματεία για τις προσπαθίες της για αυτό το ταξίδι. Πολύ ενδιαφέρον το ταξίδι ήταν αυτό. Συμφωνώ με όλα όσα είπε η κυρία Κέρ. Αλλά ήθελα να προσθέσω στην έκθεση, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ειδικότερα το κομμάτι των μεταφορών και να το διαθέσουμε και στην Επιτροπή της Τραν ε, των Μεταφορών. Γιατί πολλές συζητήσεις γίνονται και εκεί, όπου είμαι και εγώ μέλος, για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πολιτική συνοχή για την υλοποίηση των ε, έργων υποδομών. Και εκεί βλέπουμε ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα με τον υπόγειο σιδηρόδρομο στη Σόφια, ε, ώστε να κοινοποιήσουμε, να γνωστοποιήσουμε σε όλους ό,τι μάθαμε εκεί πέρα και στην Επιτροπή Τραν. Θα ήθελα εγώ να είμαι πρέσβης αυτού του μηνύματος. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Αν μου επιτρέπετε θα πω και εγώ δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία να ευχαριστήσω επίση και όλους τους συναδέλφους που ήρθαν στη Βουλγαρία. Δεν ήταν κάτι εύκολο. Είχαμε, πέσαμε σε καταιγίδα με το αεροπλάνο, έκανε τρομακτικό κρύο κατά την επίσκεψή μας, αλλά ευχαριστώ για την προσοχή σας και για τη συμμετοχή σας σε όλους τους διαλόγους. Ήταν πολύ σημαντικό. Κάναμε συναντήσει ξεκινώντας από τον Πρωθυπουργό μέχρι του εκπροσώπους των τοπικών αρχών και των διαχειριστικών αρχών ε, πολλών από τα επιχειρησιακά προγράμματα. Είχαμε επικοδομητικό διάλογο την τελευταία μέρα για την υλοποίηση της ε, τρέχουσας προγραμματικής περίοδου και είχαμε και την ευκαιρία να δούμε κάποια άριστα παραδείγματα ε, χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων στη Βουλγαρία. Κάτι νέο για τη χώρα μας. Ήταν πολύ σημαντικό λοιπόν που μας τα έδειξαν αυτά ε, και δείξαμε και την έγκριση των μελών του Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι και οι δύο, αντιπροσωπ... οι δύο επισκέψεις αυτές ήταν πολύ σημαντικές για την Επιτροπή μας, διότι οι δύο αυτές χώρες είναι από εκείνες ε, που σχετίζονται στενά ε, με την στήριξη της πολιτικής συνοχής. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε Πώ λειτουργεί επιτόπου η πολιτική συνοχή σε διάφορε περιφέρειες, σε διάφορα κράτη-μέλη, ε, που φυσικά αντιμετωπίζουν και διαφορετικά προβλήματα. Ελπίζω ότι αυτό θα μας βοηθήσει στις εργασίες μας ε, και ειδικότερα ε, στις εργασίες μας για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, ευχαριστούμε πολύ. Αναμένουμε και την έκθεση της Βουλγαρίας. Έχουμε ήδη την έκθεση της Ρωμανίας, έτσι δεν είναι. Ναι, την έχουμε στα εγγραφά μας. Και τώρα επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή διακοπή, ε, μια μικρή αλλαγή στην ημερήσια διάταξή μας. Χθες αποφασίστηκε, έκανε το ερώτημα κατά την εγκρίση της ημερήσιας διάταξης ο κ. Βανής Τελρόι. Θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους από την Ελλάδα για να μας εξηγήσουν την κατάσταση μετά από τις πλημμύρες στην Ελλάδα. Δεν θα κάνουμε συζήτηση. Θα έχουμε την επιλογή να το συζητήσουμε αργότερα σήμερα στη συνάντηση των συντονιστών. Εκεί θα συζητήσουμε κατά πόσο είναι δυνατόν να ε, εκπονήσουμε μια προφορική ερώτηση για τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Δίνω το λόγο στον κύριο Παπαδημούλη και στην κυρία Σπυράκη και παρακαλώ τηρήστε το χρόνο διότι είναι πολύ στενά τα χρονικά περιθώρια σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, όπως ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους για την ομόφωνη αποδοχή της πρότασης να συζητήσουμε έστω και για λίγο σήμερα στην Επιτροπή μας αυτή την πρόταση όπως ζήτησα και εγώ εκ μέρους πολιτικής μας ομάδας και η κυρία Σπυράκη και ο κύριος Βανίστερ Ρόι εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Πριν μία εβδομάδα μια τεράστια φυσική καταστροφή, μια πλημμύρα από αυτές που συμβαίνουν μια φορά στα 50 χρόνια χτύπησε την πατρίδα μου, την Ελλάδα και ιδιαίτερα την περιφέρεια Δυτικής Αττικής, μια περιοχή που ζουν φτωχά λαϊκά στρώματα. Και προκάλεσε μια ανθρώπινη τραγωδία. Θρηνούμε ήδη 22 νεκρούς και υπάρχουν τεράστιες υλικές ζημιές. Η κυβέρνηση, η ελληνική, έχει πάρει ήδη μέτρα για να στηριχτούν οι πληγέντες να ανακουφιστεί όσο το δυνατόν γίνεται ο ανθρώπινος πόνος, να αποκατασταθούν οι ζημιές και να μπουν μπροστά σε εφαρμογή μέτρα αντιπλημμυρικής θωράκισης. Και την ίδια ώρα υπάρχει και ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης από όλους τους φορείς της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό που προτείνω και ζητώ από την Επιτροπή μας είναι στους, στη των συντονιστών που θα γίνει σε λίγη ώρα όλες οι πολιτικές ομάδες να στηρίξουν μια πρόταση που κι εσείς έχετε σκοπό να καταθέσετε, να υπάρξει μια προφορική ερώτηση έτσι ώστε να συζητηθεί το θέμα στην επόμενη Ολομέλεια, στις 29 και 30 Νοεμβρίου, όπως έγινε και για τις πυρκαγιές στην Πορτογαλία και για τις πλημμύρες στην Ιταλία, να εκφραστεί αυτή η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη από τον ελληνικό λαό. Και δεύτερον, να ζητήσουμε ως Ευρωκοινοβούλιο από την Κομισιόν να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια στα πλαίσια των υπαρχόντων κανονισμών, έτσι ώστε αυτή η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη να εκφραστεί και με πρακτικό τρόπο, με υλικού πόρους και με ανθρώπινη βοήθεια, γιατί στις δύσκολες στιγμές μιας ανθρώπινης τραγωδίας έχει σημασία για κάθε λαό και για τον λαό τον ελληνικό να νιώθει έμπρακτα την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Σας ευχαριστώ.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 Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σπυράκη τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμόλου του συναδέλφου τη Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη για την τεράστια υποστήριξη ε, που παρήχαν ε, στον ελληνικό λαό, στο λαό μα. Ε, θέλω να πω λίγα λόγια μόνο γιατί ο αντιπρόεδρο μα, κύριο Παπαδημούλη, ήδη περιέγραψε την κατάσταση στην Ελλάδα. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω την τεράστια καταστροφή στην Αττική. Ψήμωση νεκρή είναι 22 και ενδέχεται να αυξηθεί ο αριθμός αυτός. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες εκτοπισθέντων, έχουν πληγεί επιχειρήσεις, έχουν σταματήσει ε, να λειτουργούν και οι ζημιές ε, είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστούν. Υπάρχουν υπο... Ε, ζημιές στις δημόσιες υποδομές, στους αγωγούς υδάτων. Πολλοί συμπολίτε μου έχουν μείνει χωρίς πρόσβαση σε πόσιμο νερό και ηλεκτρισμό οι δήμοι που έχουν πληγεί, συγκεκριμένα ε, Μάντρα και Μέγαρα που ανήκει η Νέα βρίσκονται στην Τουρκική Αττική. Και τώρα θα τα πω τα υπόλοιπα στα ελληνικά. Ρήτως εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος την πρότασή σας για προφορική ερώτηση στην επόμενη Ολομέλεια και παρακαλώ να συζητηθεί στην επόμενη Ολομέλεια στο τέλος Νοεμβρίου. Σε αυτή τη βάση θα ήθελα να συζητήσουμε επίσης το ενδεχόμενο να καλέσουμε την Κομισιόν να εξαιρεθεί η εθνική συνεισφορά από τις δαπάνες έργων που θα γίνουν στις πληγήσεις περιοχές, ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να πάρει την μεγαλύτερη δυνατή κοινοτική υποστήριξη ως μια σοβαρή ένδειξη κοινοτικής αλληλεγγύης. Επίσης, ζητώ να διερευνήσουμε όλες τις δυνατότητες για επιπλέον χρηματοδότηση της Ελλάδος πέρα από το Ταμείο Αλληλεγγύης, όπως ακριβώς έγινε και στην Ιταλία. Τρίτον, θα ήθελα να θέσω προ συζήτηση και προβληματισμό μεταξύ των συναδέλφων το ενδεχόμενο να προχωρήσουμε και να καλέσουμε την Κομισιόν να υπάρξουν αλλαγές στον κανονισμό για το Ταμείο Αλληλεγγύης έτσι ώστε σε χώρες που επί δέκα συναπτά έτη το εθνικό τους ακαθάριστο προϊόν πέφτει, τότε αυτές να αντιμετωπίζονται διαφορετικά σε περιπτώσει μεγάλων φυσικών καταστροφών. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου για τη στήριξη που δείχνουν στους Έλληνες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό μπορώ να πω είναι ότι στο πρόγραμμα της ημερησίας διατάξης της συνάντησης των συντονιστών έχει συμπεριληφθεί μια πρόταση για πιθανή προφορική ερώτηση και για συζήτηση στην Ολομέλεια. Ωστόσο πρέπει να αναφέρω ότι η παρούσα Επιτροπή αποφάσισε με πλήρη έγκριση της Ολομέλειας ότι όλα τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μερίδιο των διαρθρωτικών ταμείων για αποκατάσταση μετά από φυσική καταστροφή. Αυτή είναι η απόφασή μας και αναμένουμε η ελληνική κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει αυτή την επιλογή η οποία είναι ανοιχτή για όλα τα κράτη-μέλη. Ελπίζω λοιπόν να βρεθεί μια λύση. Έχετε την πλήρη συμπαράστασή μου στον ελληνικό λαό, στο, ε, στους ανθρώπους της Αθήνας. Λυπούμαστε πάρα πολύ για τις ζωές που χάθηκαν και τις υλικές ζημιές και ελπίζουμε ότι η Ελλάδα θα καταφέρει να ανακάμψει από αυτή την τραγουδία. Συνεχίζουμε τώρα με την ψηφοφορία. Ζητώ συγγνώμη. Absolutely. Let me, let me explain you. Συγγνώμη να σας εξηγήσω, λέει η Πρόεδρος. Η, μόνη διαφορά μεταξύ εσάς και των συναδέλφων που ήδη μίλησαν είναι ότι το ανέφεραν, όπου έστειλαν μηνύματα ετήθηκαν να πάρουν τον λόγο, συζήτησαν με όλες τις πολιτικές ομάδες και ζήτησαν το χρόνο αυτό. Γι' αυτό το λόγο έδωσα το λόγο σε αυτούς και τώρα σας δίνω το λόγο. Έχετε το λόγο. Σας δίνω το λόγο, εάν με ακούτε. Στροφές από τις πλημμύρες της Δυτικής Αττικής στη χώρα μου, στην Ελλάδα, που κόστησαν 21 ανθρώπινες ζωές μέχρι σήμερα 22 και τεράστιε καταστροφέ εργατικών λαϊκών οικοκυριών, αφήνοντας άστεγους χιλιάδες συνιστούν συνέπεια ενό διαχρονικού εγκλήματο. και είναι υπεύθυνη η πολιτική όλων των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την περιφερειακή τοπική διοίκηση. Η ελληνική κυβέρνηση με τι ανακοινώσει τη ξεκαθάρισε ότι δεν θα αποζημιώσει του πληγέντε σε ύψο 100% των ζημιών που υπέστησαν. Έχει αφήσει απ' έξω το πάγωμα των δανείων, την πληρωμή του έμφυα, ενώ δεν καλύπτει τι ζημιέ για αυτοκίνητα που χάθηκαν και ήταν μέσα παραγωγής για τους κατόχους τους, όπως και για βάρκε που έχασαν αλλιεί. Η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ έχει καταθέσει πριν καν τι συγκεκριμένε καταστροφέ σχετικό ψήφισμα στην Επιτροπή Ρέτζι για την άρση των απαράδεκτων περιορισμών που θέτει το Ταμείο Αλληλεγγύη, προκειμένου να αποζημιωθούν τα πληγέντα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά οι αυταπασχολούμενοι, έροντα τη σχετική απαγόρευση ότι δεν αποζημιώνονται οι ιδιώτες, όπως και για να αρθεί το απαράδεκτο όριο του 1,5% του ΑΕΠ της Περιφερειακής Ενότητας που προβλέπει το Ταμείο ως ελάχιστο όριο ζημιών. Ζητάμε να καταθέσει η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ερώτηση στην Επιτροπή για την Ολομέλεια που να συνοδεύεται από ψήφισμα με περιεχόμενο την άρση αυτών των εμποδίων βάσει του ψηφίσματος που έχει ήδη κατατεθεί από την Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στην Επιτροπή Ρέτζη. Επιπρόσθετα, να ενεργοποιηθούν κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης τόσο για αποζημιώσεις όσο και για τις αναγκαίες υποδομέ, Εκτός λοιπόν από τα μεγάλα σας λόγια περί συμπάθειας και αλληλεγγύη, εκτός και από την κουτσουρεμένη συζήτηση που δεν έγινε καν συζήτηση σήμερα, ε, καλούμε να γίνει συζήτηση και στην Ολομέλεια και να πάρθουν συγκεκριμένε αποφάσει. Η στάση σα απέναντι στο ψήφισμα του ΚΚΕ θα αποκαλύψει τι πραγματικέ προθέσει σα για το αν σκοπεύετε πραγματικά να ανακουφίσετε εργατικά λαϊκά οικοκυριά, του αυταπασχολούμενου που έχασαν το βιό του. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Επαναλαμβάνω ότι οι συντονιστές της Επιτροπής μας θα συζητήσουν σήμερα την ε, επιλογή αυτή, τη ενδεχόμενο προφορικής ερώτησης που θα συζητηθεί στην Ολομέλεια και έχουμε ήδη εκφράσει όλοι μας την υποστήριξή μας προς τους Έλληνες πολίτες. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα νομικά μέσα που υπάρχουν ώστε να υποστηρίξουμε τους πολίτες της Αθήνας και τους πολίτες των περιοχών που επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή. Έχετε όλοι μας τη συμπαράσταση για τους Έλληνες πολίτες. Συνεχίζουμε τώρα με την ημερήσια διαταξή μας και περνάμε στις ψηφοφορίες. Θα ξεκινήσουμε με την έκθεση του κυρίου Κοντζολίνο «Υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η κυρία Μπρέσο ήθελε να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Κοντζολίνου. Είχε κάτι επίγον και χρειάστηκε να φύγει και απλά ήθελε να ζητήσει συγγνώμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε στην ψηφοφορία, ξεκινώντας ε, αμέσως με την τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 53 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην NV48 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές. Πρέπει να ψηφίσουμε όλες τις έμβεις, ζητά συγγνώμη η Πρόεδρος. Πρέπει να ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες ε, της έμβη. Έμβη 50 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έμβη 52 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έμβη 53 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. NV56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εφόσον εγκριθεί καταπίπτουν οι επόμενες και πάμε στη συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην ε, τροπολογία Τη ΕΝΒΗ αριθμός 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΕΝΒΗ 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική, ε, συγγνώμη, τροπολογία 28 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ενβι 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην NV21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. NV18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. NV25 υπέρ κατά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 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 18, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 112, συγγνώμη, 117. Τροπολογία 117 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 118 υπέρ, κατά, Συγγνώμη, προφορική ερώτηση. Προφορική τροπολογία. Υπάρχει κάποια ένσταση για την προφορική τροπολογία. Όχι. Οπότε ψηφίζουμε με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 135 υπέρ, κα, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 143 υπέρ. Σωστά. 143 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 147 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 26 Πάμε κατευθείαν στην συμβαστική 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 153 υπέρ, κατά με την προφορική τροπολογία, συγγνώμη, ενστάσεις, όχι. Ψηφίζουμε την 153 μαζί με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική, ε, συγγνώμη, τροπολογία 1 των ιδιωτικών σκέψεων ε, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 27 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 με προφορική τροπολογία ενστάσεις. Όχι. Ψηφίζουμε μαζί με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην NV5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε επί του συνόλου της έκθεσης ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας και εγκρίνεται η έκθεση. Συγχαρητήρια για τον κύριο Κοτσολίνο. Ευχαριστούμε. Uh, the next... Επόμενη ψηφοφορία. Ονομοδότηση του κύριου Χέτμαν για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι η έκθεση. Θέλετε να πείτε κύριε Χέτμαν κάτι, όχι, ευχαριστούμε. Περνάμε λοιπόν απευθεία στην ψηφοφορία. Συμβιβαστική 15. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 98. Ψήφι υπέρ. ΑΕΑ 98 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 18 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 102 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 103 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 104. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται να ελέγξουμε όμως καλύτερα. Άρχεται ο ηλεκτρονικός έλεγχος. 104. Πέρας. And it is... Απορρίφθηκε πράγματι. Τροπολογία 105. Ψήφι περ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβεβαστική 19. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 108. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 109. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβεβαστική 20. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 114, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 21, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 22, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 125, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Τροπολογία 126. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβεβαστική 23. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβεβαστική 24. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 135. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 136 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το 137 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 25 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 141 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 26 ψήφι υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 144. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Τροπολογία 144. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 145. Ψήφι υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 146, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε. 146 ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίφθηκε. 147. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 148. Ψήφι υπέρ. Όχι, καταπίπτει γιατί ενεκρίθη 149 απορρίφθηκε. Όχι. Ψηφίζουμε την 148 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 150 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 151 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 152 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 158 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 159 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 160 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. The Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Με μία ψήφο διαφορά. Το 162. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 13, ψήφι περ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 163, ψήφι περ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 164. Έχει αποσυρθεί. Πηγαίνουμε στη συμβιβαστική 28. Ψήφι περ. Κατά, άποχες. Να ελέγξουμε τη συμβαστική 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, όχι. Συγγνώμη. Τέλος πάντων, έληξε η ψηφοφορία. Λυπούμε. Όχι, διακόπτουμε και ξαναρχίζουμε. Επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία επί της συμβαστικής 28. Λόγω τεχνικού σφάλματος κλείσαμε πολύ νωρίς τη ψηφοφορία. Λοιπόν, συμβαστική 28 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Τώρα λίγη ψηφοφορία. Απορρίφθηκε η τροπολογία αυτή. Που σημαίνει ότι θα ψηφίσουμε τις δύο διαγραφές. Ψηφίζουμε πρώτα απ' όλα την τροπολογία 165, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται και τώρα τροπολογία 166. Είναι διαγραφή, αλλά δεν τη ψηφίζουμε. Πηγαίνουμε στην τροπολογία 14. 14. Γιατί δεν πέρασε η συμπιβαστική. άρα ψηφίζουμε το κείμενο. Τροπολογία 14, ψήφι περ Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε, να ελέγξουμε τη 14 ή ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 167. Ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 168. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται. Συμβιβαστική 29. Θέλετε να ελέγξουμε την 168. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. 168. Πέρας ψηφοφορίας. Έγινε δεκτή με μία ψήφο διαφορά. Ευχαριστώ. Λέει κάποιος παρακαλώ λέει πρόεδρος. Συμβιβαστική 29. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 171. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 172 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 173 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτη. 175 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 177 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 178 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 179 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 180 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 30 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 184, 184 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε την τροπολογία 184, την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας, απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 31, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 32. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 190. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται. Τροπολογία 191. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 192. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 193 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 194 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 195 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 196 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 197 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 198 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Οι 190 ήταν ταυτόσιμοι. Με την προηγούμενη απορρίφθηκε και αυτή λοιπόν. Η 200 δεν καταπίπτει, είχε απορριφθεί η 191. Λοιπόν, 200 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 201 υπέρ, κατά, αποχές, γκριντ. 202 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 203 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 204 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 205 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 206 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 207 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 208 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 37 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά αποχές. Να σηκώνετε τα χέρια σας. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Να ελέγξουν. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά 17 τη ψηφοφορία. They Ζήτησα τον έλεγχο. The check Οι σύμβουλοι να μην ζητάνε, γιατί έχω αυτιά και ακούω. Δεν είναι πρώτη φορά, τελευταία φορά, να ακούμε κάποιο σύμβουλο να ζητά έλεγχο. Εσείς βεβαίως και έχετε δικαίωμα. Όχι ο συμβουλός σας όμως. Right. Απολύτως δίκιο έχετε. Δεν δέχομαι να εκφράζουν επιθυμία για έλεγχο οι συνεργάτες, οι σύμβουλοι. Τα μέλη της Επιτροπής Ρέτζι, ναι. Παρακαλώ να σιωπούν οι σύμβουλοι στη διάρκεια της ψηφοφορίας. Λυπούμε πολύ. Λυπούμε πολύ γι' αυτό. Παρακαλώ, να το προσέξουμε αυτό. Πάντως θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 19, ε, 17 λόγω αιτήματο του ΕΛΚ. Άρχεται η ψηφοφορία 17. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2.10. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 2.11. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 2.12. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Απολογία 2.17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίφθηκε. 18 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 219 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 225 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 226 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 227 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 230 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 231 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε Ελέγχουμε τη 231 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. 231. 231. The vote is closed and it is rejected. Thank you. It is rejected. Απορρίπτεται. 232 υπέρ Μπορούμε να δείξουμε τα αποτελέσματα παρακαλώ. Έξι ψήφισαν υπέρ, 30 κατά και μηδενικές αποχές. Συγγνώμη, πήγαμε πολύ γρήγορα. Προσπαθώ να μιλάω με ταχύτητα και δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, 2.32 επαναλαμβάνω. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απερίφη. 2.33 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 2.34 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 2.35 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 2.36 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 2.37 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 2.38 υπέρ, κατά αποχές απερίφη. 2.39 υπέρ κατά αποχές απερίφη. 2.40 υπέρ κατά αποχές απερίφη. Θεολογικές σκέψεις 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 21 υπέρ κατά αποχές απερίφη. Θέλετε να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 21. Είναι σαφής η έκβαση, αλλά εν πάση περιπτώσει το ελέγχουμε. Ηλεκτρονική ψήφος για την 21. Πέρα στις ψηφοφορίες βλέπετε το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Συμβιβαστική 1. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ, ποιοι είναι κατά, αποχές, Δεκτή. Συμβιβαστική υπαριθμών 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή 45 υπέρ κατά αποχές απερίφη. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 51 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 56 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 59 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απερίφθη. Ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν για την 59. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζεται. Πέρα της ψηφοφορίας. Απερίφθη πράγματι. Συμβιβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 65 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 65. Ψηφίζεται. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτή. Συγγνώμη έκανα λάθος. Συμβιβαστική 13. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Λοιπόν, συμβιβαστική 12 λέει. Πρόεδρος υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τώρα συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 36 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 71 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 72 είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 73 Κάποιος έχει ζητήσει να υπάρξει κατά διέρεση ψήφος εδώ σε δύο τμήματα. Λοιπόν, το πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα της 73 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι γίνεται και το δεύτερο τμήμα δεκτό θέλετε να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν δεύτερο τμήμα της 73 ψηφίζετε. πέρα στις ψηφοφορίες απερίφθη 74. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφη. 75. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 80 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 81 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 82 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 83 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 84 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 85 υπέρ κατά αποχές απερίφη 86 υπέρ κατά αποχές απερίφη 87 υπέρ κατά αποχές δεκτή και τώρα τελική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία Πέρα στις ψηφοφορίες, Η γνωμοδότηση λοιπόν γίνεται δεκτή. Έχουμε καθυστερήσει συνάδελφοι. έχουμε καθυστερήσει ιδιαίτερα θα έλεγα και στα πλαίσια της ανταλλαγής απόψεων με τον Επίτροπο Έτιγκερ. Θα ήθελα να σας προτείνω να ζητήσουμε από τον Επίτροπο Έτιγκερ να έρθει εδώ γιατί και αυτός έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις και αμέσως μετά θα ψηφίσουμε την έκθεση Μάλετιτς. Εντάξει, σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Θα δίνουμε το λόγο λοιπόν στον Επίτροπο Έτιγκερ. Dear colleagues, allow me to introduce you uh, and welcome on behalf of the whole Regi Committee the Commissioner Jottinger to our meeting. It was, please, can I ask you... Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω τον κύριο Έτιγκερ στη συνεδρίασή μας. Παρακαλώ να μην φωνασκείτε θα ήθελα να σας παρακαλέσω οι συζητήσεις να λάβουν χώρα εκτός της αίθουσα συνεδριάσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σας πω ότι ήταν πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας να συναντήσουμε τον Επίτροπο Έτιγκερ διότι εδώ συζητάμε το μέλλον της πολιτικής συνοχής, το χρονοδιάγραμμα του χρηματοοικονομικού πλαισίου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάμε πολλά θέματα που απτώνται του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπρεπε λοιπόν οπωσδήποτε να καλέσουμε εδώ τον Επίτροπο Έτιγκερ. Ευχαριστούμε που μα αφιερώνετε λίγο χρόνο ε, για αυτή την παρουσίαση. Ξέρω ότι είστε πολύ άσχολο και θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές κυρίες και κύριοι, Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω με την ε, Επιτροπή σας ε, για την περαιτέρω εξέλιξη της ε, δημοσιονομικής μας στρατηγικής. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα όχι μόνο άπαξ και για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σήμερα να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, αλλά να εκμεταλλευτώ και το προσεχές διάστημα ώστε να συνομιλήσω μαζί σας για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει και στις ε, πολιτικές ομάδες. Επίσης, ε, ε, σας είπα και για το... Μάλλον το Σάββατο στις 4 με την Επιτροπή Προϋπολογισμών και το Συμβούλιο συμφωνήσαμε σε ό,τι αφορά το πολιετές για τις ε, πληρωμές ε, θέλουμε να έχουμε αρκετό περιθώριο ώστε όλες ε, τις πληρωμές να μπορέσουμε να τις εξασφαλίσουμε για την συνοχή. Βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα ότι ο προϋπολογισμός και το δημοσιομικό πλαίσιο μέχρι το 2020 συμφωνήθηκε τελευταία στιγμή, δηλαδή το Δεκέμβριο του 2013. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και σιγά σιγά άρχισε να προχωρά το πράγμα. Δηλαδή σημειώθηκαν τεράστιες καθυστερήσεις ε, σε ό,τι αφορά ε, την εκταμεύση των κονδυλίων. Και για το 2017 έγινε ένας διορθωτικός προϋπολογισμός ε, για πολλά δις τα οποία δεν χρειαστήκαμε και τα γυρίσαμε πίσω. Πολύ σημαντικό επίσης ήταν και το θέμα του τι θα κάνουμε για τα επόμενα χρόνια με την άκουση του προπολογισμού για το 2013-2014-2015 είδαμε ε, να υπάρχει ανάπτυξη και οι εξελίξεις που είδαμε δεν πρέπει να επαναληφθούν. Ε, σίγουρα δεν είναι η κατάσταση ίδια, αλλά δεν θέλουμε να επαναληφθεί αυτό που έγινε το 2013-2014-2015, το 2020-2021, γιατί εκεί να δείτε καθυστερήσεις που θα έχουμε και προβλήματα. Επομένως, ήδη προετοιμάζουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020 Έχετε, φαντάζομαι, λάβει γνώση το εγγράφου προβληματισμού. Εκεί έχουμε θέσει διάφορα ζητήματα, έχουμε αναφέρει τα προβλήματα για το δημοσιονομικό πλαίσιο ε, της επόμενης δεκαετίας ε, έχουμε ε, δύο πολύ σημαντικά κενά, δύο σημαντικές τρύπες. Η μία έχει να κάνει με τα έσοδα, επειδή θα φύγουν οι Βρετανοί. Αυτό ε, μας αφήνει σε μια μεταβατική φάση, τη φάση της διαπραγμάτευσης ε, και έχουμε 10 ε, έως 12 ή 12 έως 14 δις ευρώ τρύπα ετησίως. Και έχουμε και από την πλευρά των δαπανών ένα κενό, μια τρύπα, γιατί στο Κοινοβούλιο έχετε αναλάβει νέα καθήκοντα τα οποία είτε καθόλου είτε ε, εν μέρη ε, ε, λήφθηκαν υπόψη μόνο στο πλαίσιο της δομής του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Δηλαδή έχουμε τα μεταναστευτικά ζητήματα, τους πρόσφυγες, την, τον έλεγχο των συνόρων, την προστασία των συνόρων. Έχουμε την ενίσχυση της αναπτυξιακής βοήθειας η παροχή βοήθειας για τους ε, πρόσφυγες στην Τουρκία ή ε, το θέμα της ε, έρευνας στον τομέα της άμυνας και της άμυνας γενικώ. Αν λοιπόν δούμε αυτά τα κενά και αν θέλουμε να κλείσουμε τις τρύπες αυτές στον προπολογισμό, χρειαζόμαστε μια στρατηγική και χρειαζόμαστε και πραγματικά εντατική διαπραγμάτευση και διαβούλευση το θέμα είναι πώς θα κλείσουμε ε, την τρύπα του Brexit ε, με ε, μεταφορές πιστώσεων και εξοικονόμηση 15% στον υφιστάμενο προπολογισμό, μάλλον 50% αυτά τα δύο και 50% νοπό χρήμα. Το δεύτερο κενό που είναι οι νέες δαπάνες λόγω των νέων καθηκόντων. Εδώ πρέπει τα κράτη-μέλη να επιβαρυνθούν. Γι' αυτό λοιπόν τουλάχιστον θα έλεγα το 80% των απαραίτητων δαπανών αυτών να γίνουν με fresh money, με νοπό χρήμα και 20% το μέγιστο ποσό ε, των μεταφορών πιστώσεων στον τομέα αυτό. Και έχουμε και τις αξιολογήσεις ε, που εκκρεμούν. Βλέπουμε τα προγράμματα, τα αξιολογούμε, προσπαθούμε να δούμε πού μπορούμε να είμαστε καλύτεροι, πού ε, θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες εξοικονομήσεις, πού μπορούμε να έχουμε απλούστευση κανόνων, πού μπορούμε να συγχωνεύσουμε κάποια προγράμματα για τα επόμενα χρόνια ε, αν δεν υπάρχει συνεκτικότητα ε, και όλα αυτά είναι μια προεργασία ε, για την πρόταση που θα υποβάλουμε το Μάιο του χρόνου, το Μάιο του 2018 στο Κοινοβούλιο σας. Εγώ πραγματικά είμαι υπέρμαχος της πολιτικής συνοχής, είμαι πεπισμένος για την αξία της πολιτικής συνοχής. και αν διαβάσετε και το έγγραφο προβληματισμού θα, θα δείτε τις απόψεις μας. Πιστεύω ότι για την επόμενη δεκαετία οι πολιτικές συνοχές θα δραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο ε, στην ευρωπαϊκή δημοσιονομική και περιφερειακή πολιτική. Τουλάχιστον αυτό οφείλει να πράξει. Και γι' αυτό ε, πρέπει να πω ότι σημειώνουμε κάποια πρόοδο δεν μπορούμε να διακόψουμε αυτή την πρόοδο, αυτή την πολιτική συνοχή, γιατί αυτό θέτει και σε κίνδυνο και επαμφισβήτηση και την μέχρι τώρα επιτελεστήσα ε, πρόοδο. Δεν ξέρω αν θα χρειάζεται μέχρι το 2050 η πολιτική συνοχή. Αυτό που ξέρω όμως είναι, και το λέω από τη δική μου εμπειρία, από τη δική μου την πατρίδα, ότι ξεκινήσαμε το 1990 με μια εθνική στρατηγική συνοχή στη Γερμανία για την ανοικοδόμηση της Ανατολικής Γερμανίας, ε, για ε, την εξισορρόπηση, την ισοσκέληση των δύο ε, Γερμανιών που συνενώθηκαν σε μία. Πετύχαμε. Ο Χέλμουτ Κόλ το είχε υποσχεθεί και υπήρχαν ε, πρόδι πραγματικά πάρα πολύ στο Χάλε, στην Γένα, στην Τρέσδη, στο Πότσνταμ, στο Ανατολικό Βερολίνο, στο Γκέρλιτς. Πραγματικά το Γκέρλιτς για μένα ε, είναι η ευρωπαϊκή πόλη αν θέλετε. Είναι ανατολικά της Αξονίας ε, σε μια μεθοριακή περιοχή στα όρια του ψυχρού πολέμου και από το 1990 ακολουθήσαμε μια νέα οδό, ανεξαρτησία από τη Μόσχα. Αλλά 13 χρόνια δεν ήμασταν στην Ένωση και τώρα είμαστε 13 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει ότι ο Γκέρλιτς ε, ε, ανήκει ε, και ένα κομμάτι του στην Πολωνία. Έζησε για πολλά χρόνια χωρίς την πολιτική συνοχή, 13 χρόνια είναι με, πολιτική, με προγράμματα της πολιτικής συνοχής και για τα επόμενα τουλάχιστον 10-13 χρόνια θα χρειαστεί ε, η πολιτική συνοχή στην περιοχή αυτή. Σίγουρα η πολιτική συνοχή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Χρειαζόμαστε αύξηση των κονδυλίων. Αλλά το θέμα είναι τι μπορούμε να υποστηρίξουμε. Αυτό που μπορούμε να υποστηρίξουμε είναι μικρές περικόπες στον προπολογισμό και όχι μια τεράστια αύξηση στον προπολογισμό, με το στόχο όμως η πολιτική συνεχίζει να πληγεί το λιγότερο δυνατόν από αυτές τις περικοπές. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο είναι σαφές ότι θα υπάρξουν ε, αντιθέσεις και διαφωνίες. Δεν είναι κανένα δυο, είναι 6, 7, 8 κράτη-μέλη ε, αυτά τα οποία διαφωνούν και θέλουν το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο ε, να ε, μην περιβεί το 1% στα έσοδα σε σχέση με το ΑΕΠΑ. 1% να είναι το ανώτατο όριο. Αυτό σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια. 1%. Δεν θα μπορέσουμε με 1% να χρηματοδοτήσουμε αυτά που έχουμε να επιτελέσουμε ως καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας το λέω ανοιχτά έχουμε ε, αυτά τα κράτη-μέλη που θέλουν ε, better spending, όπως λένε. Αυτό είναι το σλόγγαν. Παρακαλώ, αν ανήκετε σε αυτά τα κράτη, ασκήσετε παρακαλώ πίεση ε, να έχουμε κάτι παραπάνω από το 1%. Χρειάζεται 1% και παραπάνω για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα νέα καθήκοντα. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε στα παλαιά επίπεδα. Αυτό είναι το worst case σενάριο. Το χειρότερο σενάριο έχουμε την άμυνα, έχουμε τη μετανάστευση. Δεν μπορούμε σε βάρος πολιτικής συνοχής να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα νέα καθήκοντα. Επίσης, η ένταξη των προσφύγων πρέπει να την ε, ε, χρηματοδοτήσουμε. Και εάν τη χρηματοδοτήσουμε σε βάρος της συνοχής, έχουμε διχασμό, έχουμε διαίρεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τη Σουηδία, τη Δανία, ε, την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Γερμανία, που είναι υπέρ του δόγματος του better spending. Και απ' την άλλη έχουμε τις χώρες που δέχονται όλους αυτούς τους πρόσφυγες. Λοιπόν, χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να επιτελέσουμε τα νέα καθήκοντα ένα προπλησμό πάνω από το 1%. Υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Αν κάνουμε μια περικοπή στην πολιτική συνήθεια, 30%. Τι θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν είναι αναγκαίο. Μπορεί να υπάρχει όμως μία μείωση 10, 12, 13%. Επίσης, βλέπω μέχρι στιγμής ε, και ακούω μια άποψη ότι η πολιτική συνοχή ε, είναι κάτι που πρέπει να αποτελέσει μια προσφορά προς όλα τα κρατημέλη και προς όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, συνομιλητές μόνο τις λίγες ανεπτυγμένες ε, περιφέρειες γιατί δεν θα υπάρξει αποδοχή από τις υπόλοιπες περιφέρειες οι οποίες δεν θα μπορούν πλέον να συμμετέχουν ε, στα προγράμματα συνοχής και αυτό καταστρέφει και την όλη ιδέα της συνοχής. Άρα, ένα είναι το πολύ σημαντικό που θέλω να πω. Added value, προσθέμενη αξία. Εγώ θέλω μαζί με εσάς, που έχετε πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από εμένα, να προωθήσουμε την προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής Κάτι που το βλέπουμε στι περιφέρειε και μεταξύ των περιφερειών. Πρέπει να την αποδείξουμε, να την τεκμηριώσουμε και να την προβάλλουμε την προστιθέμενη αξία. Έχουμε διασυνοριακά προγράμματα. Γι' αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα. Στι ε, υποδομέ. Έχουμε 3, 4, 5, 6 κράτη που αφορούν ε, αυτά τα σχέδια υποδομών. Κανένα πρόβλημα. Connecting Europe, κανένα πρόβλημα. Σας ρωτώ το εξή και είναι μια ερώτηση, πρόκληση. Αν για παράδειγμα, ε, για την πολιτική συνοχή. Στη Βουλγαρία έχουμε μια συνδρομική σύνδεση. Ε, Δημόσιε συγκοινωνίε. Από τη Σόφια στην Ήπεθρο. Θέλουμε να το συγχρηματοδοτήσουμε με τα κονδύλια συνοχή. Αυτό τι είναι, είναι προστέμενη αξία. Η δημοσιονομική πολιτική θα μπορούσε να πει η Βουλγαρία μπορεί να το κάνει μόνη της αυτό. Ναι και όχι είναι απάντηση από νομική πλευρά, αμυγό, ναι. Από δημοσιονομική πλευρά, αμυγό, όχι. Δεν μπορεί να το καταφέρει η Βουλγαρία από μόνη τη. Και εγώ το λέω. Το λέω ξεκάθαρα. Ότι θέλουμε να έχουμε μια ευφυή ένωση μεταφορών ε, πιστώσεων. Αλλά και αυτό είναι επικίνδυνο και θα έρθω σε αυτό. Εγώ το πιστεύω και το εννοώ. Το ΕΠ κατά κεφαλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά μέσο όρο είναι 30.000 ευρώ. Λουξεμβούργο είναι 90.000 ευρώ. Στη Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία είναι 42-43.000 ευρώ. Στη Βουλγαρία 6.500. 6.500-90.000. Και αυτό, εάν παραμείνει έτσι, αυτό το χάσμα καταρακώνει την ευρωπαϊκή ιδέα, τα ευρωπαϊκά ιδεώδια καταστρέφει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αυτή τη διαφορά, αυτό το χάσμα, την ψαλίδα πρέπει να τη μειώσουμε. Όχι φέρνοντα προ τα κάτω το Λουξεμβούργο, αλλά ανεβάζοντα τη Βουλγαρία. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Υπάρχουν ε, κράτη, ε, να σας πω, Ρουμανία, Εσθονία, Λετωνία, Λιθουανία, οι χώρες αυτές θα μπορούσαν να πω και άλλες. Τα 13 χρόνια που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω των ενισχύσεων από την πολιτική συνοχή και από άλλα ευρωπαϊκά μέσα έχουν καταφέρει να ενισχύσουν την οικονομική τους ανταγωνιστικότητα και το κατακεφαλήν έπα. Έχει ανεβεί σημαντικά. Και αυτή τη διαδικασία πρέπει να την συνεχίσουμε και την επόμενη δεκαετία. Τουλάχιστον την επόμενη δεκαετία. Αυτό το θεωρώ απαραίτητο. Και γι' αυτό η Βουλγαρία, για παράδειγμα, χρειάζεται τα κονδύλια της συνοχής και η προστέμενη αξία έγκυται και σε ε, έργα τα οποία μπορεί να μην περιορίζονται μόνο εντός. Εγώ θα προσπαθήσω τα επόμενα χρόνια να πείσω το Συμβούλιο να μας δώσει τα μέσα για να πετύχουμε αυτή την προσθέμενη αξία. Μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Για να υπάρχουν πιο αποτελεσματικές επενδύσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα τελευταίο. Εάν κάνουμε business as usual, τότε το δημοσιονομικό πλαίσιο και τα προγράμματα ε, θα, για τη συνοχή θα αποφασιστούν το 2020. Πάλι πολύ αργά, πάλι με μεγάλη καθυστέρηση. Πάλι θα έχει χαθεί ένα έτος, στην προκειμένη προς το 2021. Δεν μπορούμε να χάσουμε άλλον ένα χρόνο. Πρέπει να μάθουμε από τα μαθήματα και από τα λάθη του παρελθόντος. Και ένα μόνο το χρονοδιάγραμμα που σημαίνει ήδη από το Μάιο του χρόνου η Κομισιόν λαμβάνει υπόψη και το Brexit και αξιολογεί και τη διαδικασία της Λευκής ε, Βίβλου και καταθέτει πρόταση για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Και την ίδια μέρα ξεκινάει η δουλειά. Και το Συμβούλιο παράλληλα ε, πρέπει να είναι έτοιμο. Με τη Βουλγαρική, την Αυστριακή και την Ρουμανική Προεδρία έχω στενές επαφές και θα έχω στενές επαφές και ενδεχομένως πριν το Μάιο του 2019, ε, μετά από ένα χρόνο δηλαδή διαβούλευση, θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε τις διαβουλεύσεις για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Οπότε θα είναι σαφές για όλους. Ερευνητές, πανεπιστήμια, δήμοι, κοινότητες, αγορά εργασίας, βιομηχανία, όλοι θα έχουν σαφή εικόνα και αυτό δείχνει χρηστή διακυβέρνηση. Φεύγουν οι φίλοι μας οι Βρετανοί και ταυτόχρονα έχουμε το πολύπλοκο, άκρος ε, πολύπλοκο ζήτημα ε, που πρέπει να μας απασχολήσει. Ε, πώς θα συμφωνήσουμε για το δημοσιονομικό πλαίσιο της επόμενης δεκαετίας. Δυστυχώ, επειδή στι 11 έχω μια διάσκεψη που πρέπει να προεδρεύσω, στι 11 παρα 10 πρέπει να φύγω. Όμω ε, είμαι έτοιμο να ξεκινήσω για να Λεβάρη, οι συνάδελφοι Κρέτσου, Τάισεν που είναι οι, ε, οι δήμονε ε, για τα θέματα τη πολιτική συνοχή θα μα βοηθήσουν και σίγουρα και η δική σα εμπειρία και η δική σα γνώση θα μα βοηθήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντική και η δική σα συμβόλη. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Βλέπετε ποιο είναι το πλαίσιο, έχετε τις πληροφορίες, ξέρετε ότι ε, έχουμε πολύ λίγο χρόνο για σήμερα, οπότε θα ζητήσω τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων να πάρουν το λόγο τώρα και να είναι πολύ σύντομη, ένα λεπτό ο καθένας, ε, λίγο παραπάνω, για να έχει τη δυνατότητα ο κ. Σατικέρ και να απαντήσει. Ε, για το έλκα. Όσοι τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας ε, αδράξουμε τη στιγμή και ας πάρουμε τις ε, πληροφορίες που μας δώσατε ως δικό μας θεματολόγιο. Γεγονός που σημαίνει ότι από τώρα θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις εργασίες μας, τις δυνατότητες που έχουμε ως Κοινοβούλιο για να δράσουμε ρεαλιστικά για τα όλα σημεία που αναφέρατε. Έχουμε τα πέντε σενάρια, αλλά αυτά που είπατε σήμερα είναι πιο συγκεκριμένα και επικυρώνουν ε, με πολλούς τρόπους ολόκληρη την ενωσιακή πολιτική συνοχής και θέτει και ορισμένα ερωτηματικά για την προστιθέμενη αξία και για τις προετοιμασίες που θα απαιτηθούν επιπλέον. Εμείς πιστεύω έχουμε ήδη βάλει τους θεμέλιους ε, λίθους για τη συζήτηση στην Ολομέλεια και αυτό που ακούσαμε χθε από τον κύριο Πρεσκά από την Κομισιόν ήταν, μας είπε ήδη καταβάλουμε προσπάθειες για μια πιο αποτελεσματική, απλουστευμένη πολιτική συνοχή στην οποία θα έχουμε εξετάσει γραμμή προς γραμμή για να δούμε τι θέλουμε για την επόμενη προγραμματική περίοδο, τι θα κρατήσουμε, τι θα παρατήσουμε. Και αυτό θα συζητήσουμε και τους επόμενους μήνες στην Επιτροπή μας. Οπότε, όπως λέτε, Εάν υπάρχει δυνατότητα με το δικό σας πλαίσιο το Μάιο ε, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Και εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο. Γιατί άκουσα αυτή τη βδομάδα την Κομισιόν η οποία λέει ότι προετοιμαζόμαστε άρθρο προς άρθρο και άκουσα και το Συμβούλιο ε, Γενικών Υποθέσεων την περασμένη εβδομάδα συμφώνησαν ε, επί του κειμένου το οποίο είχε προετοιμαστεί με σε συνεργασία με τη Μαλτέζικη Προεδρία και αν το διαβάσετε θα δείτε τα ίδια λόγια με αυτά που είπατε εσείς κύριε Επίτροπε σήμερα. Ε, επικυρώνεται η αξία της πολιτικής συνοχής. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κάποια σημεία που μας απασχολούν. Ε, ναι, δεν θέλουμε να ξανακάνουμε τα ίδια λάθη και να κρατήσουμε τα κεντρικά σημεία στο επίκεντρο της μελλοντική ε, στρατηγικής και στο μέλλον του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Έχουμε τον Γιάνν Άλμπρεχτ εδώ που κάθεται εντελώ αριστερά μου ε, και ο οποίο θα θέλει να μιλήσει ε, και μπορεί να μα βοηθήσει να επιταχύνουμε. Η κυρία Κρέλ, ε, εκ μέρου των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, με ικανοποίησε ιδιαίτερα αυτό που άκουσα από εσάς ε, και πραγματικά ε, θα σας υποστηρίξουμε. Ελπίζω να πετύχετε στις προσπάθειές σας και ελπίζω και στη δική μου χώρα να πετύχουμε να είναι διαθέσιμος περιορισμός που θα ξεπερνάει το 1% αν έχουμε ε, μέχρι το 15% περικοπές ε, της πολιτικής συνοχής, λέτε μόνο εσείς, αλλά εγώ νομίζω ότι ήδη θα είναι με το κατά πόσο μπορούμε να συνεχίσουμε να ε, έχουμε μια αποτελεσματική πολιτική συνοχή. δώσατε κι εσείς ε, πάρα πολλά ε, στοιχεία που το, νομίζω τεκμηριώνουν αυτό. Είπατε ότι ε, δεν συζητήθηκε το θέμα ενός νέου συστήματος ιδίων πόρων ε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μεταγενέστερο σημείο που θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ε, νέο σύστημα και πρέπει να σας πω ότι η δική μας επιτροπή είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε πάρα πολύ σκληρά ε, σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα που αναφέρατε, ώστε να έχουμε πριν το Μάιο του 2019 τον πρώτο τριμερή διάλογο. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι ο κανονισμός ε, για το κανονισμό για το νομικό πλαίσιο ε, θα πρέπει να έρθει πάρα πολύ νωρίς για να μπορούμε ταυτόχρονα, δηλαδή να έχουμε παράλληλα να τρέχουν διαπραγματεύσεις πολιτικής συνοχής και πολιετές. Ευχαριστώ κύριο Βαν Μίλτε Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε. Willkommen, Herr Kommissar. Θα συνεχίσω όμω τα αγγλικά. Το είπατε σαφέστατα. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα λεφτά. Τεράστια πρόκληση. Και αυτό με οδηγεί σε κάποιε παρατηρήσει σε κάποιε ερωτήσει. Πρώτα απ' όλα, θα ήμουν περίεργο να μάθω ε, για την αιρεσιμότητα, για τις αιρεσιμότητες. Τι προσέγγιση έχετε όταν λέμε ότι απαιτούνται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ε, μεγάλο σύνδεσμος με το ευρωπαϊκό εξάμενο και να ξοδέψουμε τα λεφτά έτσι ώστε να έχουμε ένα ε, ορθό ε, και καλό ε, επενδυτικό περιβάλλον. Τι γίνεται με την αρεσιμότητα. Μιλήστε για αρεσιμότητα και για το κράτος δικαίου, για τις ζαπάνες, για την πολιτική συνοχή. Οπότε η ερώτησή μου είναι μελετάτε αυτές τις ιδέες. Και η δεύτερη μου ερώτηση είναι τι θα γίνει με την αυξημένη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων. Τι ιδέες έχετε γι' αυτό πώς θα κάνουμε περισσότερα με λιγότερα λεφτά. Και οι τελευταίες δύο μου ερωτήσεις, τι γίνεται με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, αφού κάνετε διάφορες δηλώσεις και εσείς και ο κύριος Γιούνκερ ότι πρόκειται για μια πολιτική επιτροπή, ε, γιατί να μην εστιαστούμε στο να ευθυγραμμίσουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο σε μια περίοδο ενδεχομένω δύο πενταετιών ώστε να προσαρμοστεί και στη στρατηγική του 2030, τη δεκαετή, και στη στρατηγική για μετά το 2030 και για την προετοιμασία αυτής της στρατηγικής. Και μετά τι γίνεται με την απλούστευση των κονδυλίων, γιατί όχι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση να μην προσαρμοστεί στα διαρθρωτικά ας πούμε ταμεία, γιατί έχουμε τόσα πολλά διαφορετικά ταμεία που θα χρειάζεται κάποια απλούστευση. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, πρόκειται για τον συντονιστή του Άλντε. Δίνω το λόγο στον κύριο Ομαγζέ από την ΚΟΕ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για την έκκλησή σας για να διατηρηθεί η συνοχή. Βλέπω ότι δεσμεύεστε όπως και ο Πρόεδρος Γιούνκερ στη διασκέψη των Προέδρων των ε, υπερπόντιων περιοχών, περιφερειών. με διαβεβαίωσαν περισσότερο οι δηλώσεις του κ. Γιούνκερ από τις δηλώσεις του Πρόεδρου Μακρόν. Και έχετε δίκιο, το πρόβλημα σήμερα βρίσκεται στο Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν θα πρέπει να συνεργαστούν ώστε να ε, επηρεάσουν τα πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η έκκληση που κάνετε, ε, μας κάνετε μια έκκληση να μην μιλήσουμε για πάνω από ένα λεπτό, οπότε έχω μία ερώτηση για σας οι επιπτώσεις του Brexit. Μήπως τις έχουμε υπερτιμήσει λίγο. Διότι ξέρουμε ότι με τη Βρετανική έξοδο τελικά αυτό που χάνουμε δεν είναι τόσο μεγάλο ποσό. Και μήπως τελικά το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση μια οργάνωση διαχείρισης κρίσεων, κρίσεων οι οποίε εντείνονται διαρκώς, ε, το είπε ο πρόεδρος της Γαλλική Δημοκρατίας. Και τελικά απαιτούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει όλο περισσότερα με αρμοδιότητες που δεν είναι δικέ της ε, κατά προτεραιότητα. Ζητάμε συνέχεια στην Ευρώπη να υποστηρίξει πράγματα χρησιμοποιώντας αρμοδιότητες ε, και θυσιάζοντας οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις συνθήκες δείτε το άρθρο 174 που αφορά ε, την ε, κοινωνική και οικονομική συνοχή. Οπότε το ερώτημα που έχω να σας ε, θέσω είναι πώς μπορούμε να βγούμε από αυτή την αντίφαση. Και όπως είπε και η Κωνσταντς, ο πιο βέβαιος δρόμος είναι να κινηθούμε προς ιδίους πόρους για να μπορέσουμε να λάβουμε όλες αυτές τις ευθύνες, γιατί προτεραιότητες υπάρχουν παντού σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος έχετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις ωραίες ιδέες τις οποίες εκφράσατε. Συμφωνώ και με πολλά από αυτά τα οποία είπατε. Είπατε ότι θα στηρίξετε τις χώρες που δεν είναι προχωρημένες οικονομικά. Αναφερθήκατε και σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει παλιότερα στη Λιθουανία Έχω την εντύπωση ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να καταφέρουμε να βρούμε τα χρήματα τα οποία έχουμε αποφασίσει ότι χρειαζόμαστε. Θυμίζω ότι το 2019 θα έχουμε τις εκλογές, ένα νέο κοινοβούλιο, μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα θα παραπεμφθούν στο 21 και 22. Ενώ τώρα είμαστε στο 2017, έστω στο τέλος του 2017 και η χρήση των πιστώσεων αυτών βρίσκεται ακόμα στην αρκτική φάση και νομίζω ότι οι ευρωπαϊκές επενδύσεις για τις χώρες με τα μεγαλύτερα οικονομικά θέματα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι των επενδυτικών δυνατοτήτων που φτάνουν στις χώρες αυτές. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω για την Ιγναλίνα, την περίπτωση της Ιγναλίνα, τι θα γίνει. Ευχαριστώ τον Επίτροπο, λέει η κυρία Τρία σενάρια από τα πέντε έχουν μειώσεις και για την ΚΑΠ και για την πολιτική συνοχή δυστυχώς. Απαιτούνται διαφθρωτικές αλλαγές σε σχέση με το ευρωπαϊκό εξάμεινο με θετικά κίνητρα μέσα από την πολιτική της συνοχής. Η πολιτική συνοχής ε, δεν είναι τέλεια. Παρ' όλα αυτά ε, για πολλές χώρες οι μοναδικές πραγματικές επενδύσεις προέρχονται από τη συνοχή. Συνεπώς λοιπόν τα πράγματα δεν φαίνονται καλά για την συνοχή. Θα πρέπει να τη βελτιώσουμε και όχι να την αποδυναμώσουμε. Και φυσικά το θέμα της άμεσης διαχείρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επανεξεταστεί για να μην δημιουργηθούν απειλές για την ε, συνοχή σε επίπεδο περιφερειακό εδαφικό. Θα πρέπει να συμμετέχουν στην διαχείριση όλο και περισσότερο από τις περιφερειακές αρχές και σχέση με τη μακροαιρεσιμότητα και το 24 ε, υποτίθεται ότι στα πλαίσια του κανονισμού θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε το μέτρο αυτό. Θα πρέπει οι λοιπόν μεταρρυθμίσεις να μην χρηματοδοτηθούν από την πολιτική συνοχή, και να είναι μια προϋπόθεση με βάση την οποία θα πάρουν τα χρήματα οι διάφορες χώρες. Τώρα για το Ταμείο Αλληλεγγύης θα ήθελα να μάθω από τον Επίτροπο και λόγω των τραγικών συμβάντων των τελευταίο καιρό σε ορισμένες χώρες υπάρχει η δυνατότητα για αύξηση του ποσού για το Ταμείο αυτό, το Ταμείο Αλληλεγγύης ή έστω να υπάρξουν περισσότερες εξαιρέσεις για την εθνική συμμετοχή. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ομιλητέ ακόμα. Ένα λεπτό καθένα. καθένας. Η κυρία Μάλετιτς. Ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Είμαστε ευτυχείς που έχουμε σας επίτροπο για τον προϋπολογισμό γιατί κατανοείτε την περιφερειακή πολιτική. Αυτά τα οποία είπατε ήταν θετικά για την πολιτική συνοχή. Είπατε ότι μια μικρή μείωση είναι κάτι το οποίο δεν θα αποφύγουμε και θα πρέπει να φροντίσουμε να μην ε, βλάψει ουσιαστικά την πολιτική μας στον τομέα της συνοχής. Λόγω λοιπόν αυτών τα οποία είπατε, λόγω του ότι απαιτείται μια ισχυρότερη πολιτική συνοχής, δεν μπορούμε να έχουμε έναν πολυδιασπασμένο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ένας του πυλώνας ε, μέσα από τις ε, διαφθρωτικές μεταρρυθμίσεις ε, παρουσιάζει κινδύνους για την ακαιρεότητα του προϋπολογισμού αυτού γιατί μπορεί να δημιουργήσει μια πολυδιάσπαση των διαθέσιμων πιστώσεων. Σε ποιο βαθμό κάτι τέτοιο θα επηρεάσει την πολιτική αυτή. Κύριε Σαριμόντ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, μου άρεσε πολύ η ειλικρίνειά σας, τα είπατε πολύ ντόμπρα και πάντα είστε σαφεί και συγκεκριμένα στην μιλάτε για την πολιτική συνοχή. Και επειδή εκφράσατε και την ε, πίστη σας ε, στην ε, πολιτική συνοχή, θέλω να σας ευχαριστήσω. Ήταν σαφής η ομολογία σας υπέρ αυτών των αρχών. Ελπίζω και άλλοι υψηλά ιστάμενοι να κάνουν το ίδιο. Δύο ε, είπατε. έχουμε τις με τα έσοδα το κενό από το Brexit. 10 με 40 ε, και λέτε ότι πρέπει να κάνουμε και κάποια εξοικονόμηση αλλά έχουμε και το, την άλλη τρύπα με τα έξοδα, με τις δαπάνες. Στην πρώτη περίπτωση είπατε το ίμιση να είναι από εξοικονόμηση, άρα γύρω στα 20. Ε, και στο, στη δεύτερη περίπτωση το 20% είναι και αυτό κάποια δις. Πώς θα τα καταφέρουν αυτά. Αυτά ήταν οι ερωτήσεις. Πρόεδρος. Καταλάβατε κύριε Επίτροπε ότι χρειάζεται ακόμα μία συνάντηση. Γενάρη, Φλεβάρη, είπατε, ε, τέλος πάντων, αν μπορείτε τώρα, καλό είναι να μας δώσετε πάντως και κάποιες προκαταρκτικές απαντήσεις. Το Φεβρουάριο θα μπορώ να δώσω σίγουρα, κυρία Πρόεδρε, πολύ πιο συγκεκριμένες απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα και σίγουρα το Μάιο μια πολύ πιο ενδελεχή απάντηση. Προσπαθώ τώρα να απαντήσω σε σχέση με το τι γίνεται στο πλαίσιο της εργασίας μας σε επίπεδο κομισιών, ε, κρατών μελών και διαφόρων άλλων ε, φορέων και θεσμικών οργάνων. Σε ό,τι αφορά το σύστημα ιδίων ε, πόρων. Ξέρετε την έκθεση Μόντι. Εμείς ό,τι αφορά τα έσοδα θέλουμε μια διαφοροποίηση. Να έχουμε δηλαδή νέους ίδιους πόρους. Έναν, δύο ή τρεις Και θα μπορούσε να ήταν ε, πολύ έξυπνο να πούμε ότι δεχόμαστε 1% του καθάριστου εγχώριου εισοδήματος αν τα κράτη-μέλη on top βρουν δύο νέους είδους πόρους. Παραδείγματο χάρη ή ε, το, την εισφορά για το διοξίδιο, είτε φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή το ETS. Έτσι, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πούν στα κοινοβούλια ότι δεν χρειάζεται να εκταμευτούν περισσότερα κονδύλια από τους εθνικούς προπολογισμού, αλλά τα νέα καθήκοντα ε, θα χρηματοδοτούνται με πρόσθετους ίδιου πόρους. Το χρονοδιάγραμμα το οποίο σας ανέφερα ε, για να ε, τηρηθεί θα πρέπει να έχουμε σύντομα ε, και προτάσεις για το νομοθετικό πλαίσιο. Λίγες εβδομάδες θα έλεγα διαφορά από το πολιετές για να μπορέσουμε σε βάθος να έχουμε διαβουλεύσεις και να μπορέσουμε να λάβουμε αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά την αιρεσιμότητα. Πραγματικά έχουν τεθεί διάφορα ερωτήματα. Θέλουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο και η συστάση αναχώρα να είναι ε, ειδικέ αναπεριφέρειας συστάσεις μήπως και να δούμε τι προτεραιότητες ε, πρέπει να εκταμιεύσουν τα κράτη-μέλη, τι πόρους από τα να πρέπει να εκταμιεύσουν για να ε, φέρουν σε πέρα σε αυτές τις προτεραιότητες. Δεν είναι εύκολο. Θέλουμε σαφήνεια, θέλουμε ασφάλεια και για την πολιτική συνοχή για πολλά χρόνια, για έναν μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Πέντε ή και παραπάνω και για το πολιτές συνομικό επίσης. Το ρούλο βλό, το κράτος δικαίου είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό και αιρεσιμότητα. Αν ένα ε, κράτος μέλος ε, έχει κάποιες ε, ανησυχίες, ε, ε, παραδείγματος χάρη το θέμα της ανεξαρτησίας τα κτλ. Ή αν εκεί που έχουμε τις συστάσεις για το κράτος δικαίου έχουμε κάποιες εξελίξεις, έχουμε κάποια πρόοδο. Αυτό είναι ένα θετικό κίνητρο που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στα κράτη. θα μπορούσαμε να βάζουμε το 10% σε ένα κοινό κορβανά και το 1% από τα κράτη. Άρα το 10% ουσιαστικά θα ήταν κίνητρα για να σημειώσουν πρόοδο τα κράτη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Το βασικό μου πρόβλημα είναι η ομοφωνία. Την Παρασκευή και Σάββατο πρωί 4 το πρωί Θέλουμε πλειοψηφία από το Συμβούλιο, πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο. Για το πολιτέ χρειάζομαι πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, αλλά ομοφωνία στο Συμβούλιο. 27 κράτη-μέλη, 27 υπουργού οικονομικών, 27 υπουργού εξωτερικών. Ουσιαστικά 27 αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων. Συν τα εθνικά κοινοβούλια, που και αυτά πρέπει να υποστηρίξουν. Και μπορώ να σα πω, κάποια εθνικά κοινοβούλια ξέρουν και αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά τη σημασία της πολιτικής συνοχής. Αλλά δεν έχουν ασχοληθεί και τόσο με το θέμα. Γιατί έναν μόνο στόχο κάτω από το 1%. το better spending που σας είπα. Και δεν μου αρέσει αυτή η έννοια better spending. Παντού μπορεί να γίνει αυτό. Όταν πάω να αγοράσω κάτι, ένα δώρο. Ή όταν η γυναίκα μου αγοράζει καινούργια έπιπλα ή όταν ε, ανεγείρεται ε, δικό δίκτυο, ένας νέος δρόμος ε, από ένα δήμο. Παντού μπορούν να έχουμε better spending. Αν από τα 100 που παράγει ένας πορτεσέτ του παίρνουμε τα 50 για να πληρώσει φόρους ε, τις ε, κοινόχρηστες ε, κοινοφέλης πέσης και τα λοιπά. Και δίνει ένα ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες. Δεν είναι δυνατόν. Χρειάζεται όμως ομοφωνία. Πέντε Επτά, πέντε συν 5, τα χρόνια δηλαδή. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω τώρα. Γενάρη, Φλεβάρη θα μπορώ να σας δώσω περισσότερα στοιχεία. Επίσης και με τα προγράμματα έχουμε την συνοχή, έχουμε το σχέδιο Juncker, έχουμε ε, το Connecting Europe. Δεν τα έχουμε όλα ε, συμφωνήσει την ίδια στιγμή, ούτε έχουν όλα τον ίδιο χρονικό ορίζοντα. Ε, αυτό το ενίο βιβλίο, Rule Book, ε, Single Rule Book και η διαχείριση και απλούστευση, πώς θα τα πετύχουμε όλα αυτά, πώς θα τα συνδέσουμε μεταξύ τους όλα αυτά. Έχουμε τελείως διαφορετικές εντολές έχουμε και το Brexit, το λογαριασμό. Δύο λογαριασμούς. Ο ένας λογαριασμός πάει στο Λονδίνο. Μέχρι τις 29 Μαρτίου του 2019 τι πρέπει να πληρώνουν οι Βρετανοί. Και μέχρι το 2020 για το πολιετές. Και εμείς είναι ένα. Νησιν τρία, συγγνώμη. Οι υποχρεώσεις ε, και οι πληρωμές μέχρι το 2021 καινή συνεχί μετά για τις ε, συντάξεις, ε, όχι των των Ευρωπαίων. Μπορεί να ζήσουν ε, άλλα 40 χρόνια. Άρα και αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αυτό είναι ο ένα λογαριασμό. Και ο δεύτερο είναι δικό μα. Μετά τη μεταβατική μα λείπουν 10, 12, 14 δι. Αν χρειαζόμαστε ομοφωνία μπορεί να μην μπορέσουμε να έχουμε όλο αυτό το ποσό, να το καλύψουμε. Αν όμως αποχωρήσουν οι Βρετανοί, πρέπει να υπάρξουν περικοπές λένε κάποιοι. Ούτε και αυτό μου φαίνεται σωστό. Δηλαδή ούτε το ένα μπορεί να γίνει 100% ούτε το άλλο. 50-50 πρέπει να είναι. 50% οι περικοπές, 50% νοπό χρήμα. Έπειτα, έχουμε ένα άλλο θέμα. Πώς χρηματοδοτούνται τα νέα καθήκοντα χωρίς να πληγεί η πολιτική συνοχή. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για τα νέα αυτά καθήκοντα, αλλά και τα ήδη υπάρχοντα, να μπορέσουμε να τα εξυπηρετήσουμε. Αν όμως δεν έχουμε νοπό χρήμα, έχουμε ήδη την ε, ε, υποχρέωση να φέρουμε σε πέρας πρώτα τα υφιστάμενα καθήκοντα και μεταξύ αυτών πολύ μεγάλη σημασία έχει η πολιτική συνοχής. Για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όλε αυτέ τι ανάγκε, χρειάζονται χρήματα από τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάπτυξη, ε, που μπορεί να εγγραφεί στον προπολογισμό. Και αυτό δεν θα πρέπει να είναι σε βάρο τη πολιτική συνοχή διότι πρέπει να υπάρχει δημοσιονομική ε, ακρίβεια ε, και να είναι σαφή τα πράγματα. Δεν μπορούμε να έχουμε περικοπές στην Ήπεθρο, στον ορίζοντα 2020, στη συνοχή. Εγώ θεωρώ ότι χρειαζόμαστε δέκα δις για τις ε, νέε αυτέ δαπάνε που θα προκύψουν και νομίζω τα δύο από αυτά πρέπει να προκύψουν από νέο χρήμα. Για το Ιγναλίνα. Υπάρχει υποχρέωση για την αποσυναρμολόγηση. Θα πρέπει να προβλεφθεί ε, και, στον επόμενο, και στην επόμενη πρόβλεψη για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν ξέρω ακριβώς σε ποιο πρόγραμμα θα συμπεριληφθεί όμως δεν θα πρέπει να καλυφθεί μόνο από το Ταμείο Συνοχής. Δεν μπορεί να επιβαρυνθεί μόνο ο προϋπολογισμός ε, συνοχής ε, για το Ιγναλίνα. Θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα κονδύλια για την επόμενη δεκαετία που θα διατεθούν προς αυτό το σκοπό. Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, θέλω να τηρηθούν οι προθεσμίες, να μην έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς που θα συσσωρεύονται στον Περλεμό. αλλά πρέπει εμείς να είμαστε ακριβείς και συνεπείς αλλά πρώτα να έχουμε και το λογαριασμό που δείχνει ότι έχει γίνει το έργο, γιατί δεν θα πληρώνω για κάτι που δεν έχει γίνει. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ, ευχαριστούμε για την αναρκτήρια ομιλία σας, για την ειλικρίνεια με την οποία συζητήσετε μαζί, μαζί μας. Σας περιμένουμε να μας ξαναεπισκεφτείτε. Ευχαριστούμε. Thank you very much, σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Ε, καταλάβατε ότι ήταν σημαντικό να συναντήσουμε τον Επίτροπο Έρτιγκερ. Και ήταν επίσης σημαντικό να διαπραγματευτούμε μαζί του την επόμενη συνάντησή μας με την Επιτροπή μας. Θα επανέλθουμε τώρα στις ψηφοφορίες. Θα ξεκινήσουμε με την γνωμοδότηση που έχει προετοιμάσει η κυρία Μαλέτιτς, έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών για τις αιτήσιες δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κυρία Μαλέτιτς δεν θέλει το λόγο. Περνάμε λοιπόν στις ψηφοφορίες αμέσως. Ξεκινάμε με τη συμβιβαστική 1. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά, αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 2. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 3. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά, αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 4. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές δεκτή. Περνάμε τώρα στην 41. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές απερίφη 42 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απερίφη. 44 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 46 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφη. 48 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι απερίφη, αλλά στο ελέγξουμε. Η 48 ψηφίζεται, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες απερίφθη πράγματι. Συμβιβαστική 5. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Περνάμε τώρα στην προφορική τροπολογία στην 61, προφορική 1 στην τροπολογία 61. Υπάρχει μια αντίρρηση για την ψηφοφορία, όχι, ψηφίζουμε λοιπόν την προφορική τροπολογία, ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 64, ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές Λοιπόν, 64 ψηφίζουμε. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Περνάμε συνεπώς στη συμβιβαστική 6. Είναι υπέρ, κατά, αποχές. Γίνεται δεκτή η 73 μένει τώρα. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές απερίφθη. Και τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Τέλος. Δεκτή. Συγχαρητήρια κυρία Μάλετιτς. Καλώς. Τώρα έχουμε τελειώσει τις ψηφοφορίες μας για σήμερα. Θα περάσουμε για την πρώτη, στην πρώτη μάλλον ανταλλαγή απόψεων στην έκθεσή μας για την ενίσχυση της ε, οικονομικής και περιφερειακής συνοχής, 7η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση δημοσιεύθηκε στην 9η Οκτωβρίου. Είναι ένα κεντρικό έγγραφο στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων ε, της επομενης ε, προγραμματικης περιόδου. Η Επιτροπή Ρέτζι θα ξεκινήσει, αποφάσισε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας σχετική με την άποψη του Κοινοβουλίου. Ο εισηγητής μας λοιπόν θα συζητήσουμε σήμερα για πρώτη φορά τις προτάσεις του. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζουλόν για να μας παρουσιάσει τις θέσεις του και μετά θα δώσω το λόγο στους Κιώδης. η συζήτηση είναι η πρώτη ευκαιρία να σχολιάσουν την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την 7η έκθεση. Θα δώσω το λόγο και στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, κύριε Ζουλό, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ξέρουμε όλοι ότι η 7η εκθέση συνοχής είναι ένα έγγραφο εξαιρετικά σημαντικό. Παρέχει πολλά δεδομένα σε βάθος αναλύσεις για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η εκθέση όμως αυτή είναι επίσης ε, και εξαιρετικά επίκαιρη. εμφανίστε σε στρατηγική στιγμή λίγους μήνες ε, πριν γίνουν οι δημοσιονομικές και νομοθετικές προτάσεις της Κομισιόν από τους Επιτρόπους. Μας επιτρέπει λοιπόν να αποκομίσουμε κάποια διδάγματα από την πολιτική συνοχή και από τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια. Γνωρίζουμε, το είδαμε και σήμερα το πρωί, ότι υπάρχουν διάφορες απειλές, ερωτηματικά για το μέλλον ε, της πολιτικής συνοχής. Ακούσαμε τον Επίτροπο Έτιγκερ, μας είπε πολλά πράγματα ενδιαφέροντα, καθησυχαστικά σίγουρα, αλλά ανέφερε και κάποιες προοπτικές, κάποια υποθετικά σενάρια μείωσης ε, των κονδυλίων. Παρότι, όπως γνωρίζουμε όλοι, το γεγονό ότι η πολιτική συνοχή έχει αποδειχθεί αποτελεσματική και αναγκαία για όλους μας στην Ευρώπη. Τώρα για το περιεχόμενο της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λυπούμαστε, λείπουν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις για το μέλλον, παρότι δεν είναι τελική. Ε, Κάποια σημεία μου φάνηκαν πολύ ενδιαφέροντα στο έγγραφο. Καταδεικνύει κάποιε επιτυχίε αυτή τη πολιτική συνοχή για τη μείωση των ανισοτήτων σε πολλέ ευρωπαϊκέ περιφέρειε Επίση, καταδεικνύει τι προοπτικέ, τι διαπιστώσει ε, που είναι ανησυχητικέ, ε, το ποσοστό ανεργία, τα διακυβεύματα, τι επιτυχίε, ε, την πραγματική σύγκληση ανάλογα με την περιφέρεια ή τη χώρα. Ένα θέμα στο οποίο πρέπει να επανέλθουμε η έκθεση μας ε, δίνει να καταλάβουμε ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η πολιτική συνοχή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε και ο Επίτροπος είναι κάτι καλό, είναι μια πολιτική στην την οποία προσυπογράφω εγώ όπως και εσείς. Ε, είναι αισιόδοξη η έκθεση και κάνει πολύ σαφείς συστάσεις. Αναφέρει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει ένα μήνυμα και μια υλοποίηση ισχυρή ε, όσον αφορά τη ριζική ε, απλούστευση και επίσης ε, αναφέρει διάφορα θέματα που πρέπει να αναπτυχθούν το ζήτημα των ε, ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης τους θύλακες φτώχες που υπάρχουν ή που μπορεί να αναπτυχθούν σε, ορισμένα, σε ορισμένες περιοχές και μετά αναφέρει και αυτή την κατάσταση στην έκθεση ορισμένων περιφερειών που παγιδεύονται ε, η παγίδα αυτή του ενδιάμεσου εισοδήματο ε, και ε, αδυναμίας ανταγωνισμού που βρίσκονται σε δύσκολη θέση απόψη προόδου είναι ένα ζήτημα το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να ξαναδούμε. Όλα αυτά φυσικά δεν είναι όλα τα θέματα που αναφέρονται στην έκθεση Πιστεύω ότι γενικά με αυτή την έκθεση δεν πρέπει να παραμείνουμε στα λόγια, στις αναλύσεις, στις σκέψεις, στους γενικούς προβληματισμούς. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή μπορεί να μας βοηθήσει να εξάγουμε μηνύματα σαφή, καθαρά, τα οποία θα γίνουν ακουστά. Θα μπορείς να μας ανοίξει οδούς ε, ε, βελτίωσης ε, και εξέλιξης διότι ξέρουμε ότι έχουμε δεσμευτεί για αυτή την πολιτική συνοχή. Τα πράγματα προχωρούν αρκετά γρήγορα ε, στην Κομισιόν όπως είδαμε, όπως ξέρουμε ε, πολλές οδοί ήδη έχουν σχεδιαστεί το να ληφθούν υπόψη τα συμπληρωματικά κριτήρια πέραν του ΑΕΠ, η διατήρηση των εξάντε αιρεσιμότητας, της εκ των η προσέγγιση της έκθεσης με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και μετά όλα τα ζητήματα που αναφέρθηκαν για το μέλλον ε, του Κοινωνικού Ταμείου, αν θα βγει ή όχι από την πολιτική συνοχή. Ε, εγώ είμαι υπέρ μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης. Ε, πιστεύω ότι αυτό είναι κλειδί για την επιτυχία της. Το Κοινοβούλιο θα χρειαστεί να εκφέρει γνώμη για όλα αυτά τα θέματα. Εγώ θα συνεργαστώ με όλους τους κοιοδησίγητες και τους συναδέλφους για να εργαστούμε γρήγορα επικοδομητικά για το μέλλον αυτής της πολιτικής ε, συνοχής. Πράγματι το χρονοδιάγραμμα μας περιορίζει για να μπορέσουμε να χαράξουμε οδούς ε, και προτάσεις πριν από την ε, Κομισιόν. Σε κάθε περίπτωση εγώ χαίρομαι που έχω εργαστώ σε αυτό το θέμα και Πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι θα συνεργαστούμε ώστε να είναι ε, όσο το δυνατόν πιο επικοδομητικό το αποτέλεσμα αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα αλλάξω λίγο τώρα το σειρά της ε, συμμετοχής και θα σας εξηγήσω γιατί. Διότι έχουμε εδώ τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίοι έχουν προετοιμάσει κάποια παρουσίαση για την 7η ε, έκθεση συνοχής ο κύριος Νίκο Δημικέλης και ο Φίλιππος Μουφόρτ παρουσιάσουν σε ένα δεκαλέπτο την ε, άποψη της ε, Κομισιόν. Έχετε το λόγο παρακαλώ κύριε Δημικέλη. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, υπάρχουν ε, πολλές πληροφορίες στην έκθεση αυτή και γι' αυτό θα συγκεντρώσω την προσοχή μου σε τέσσερα θέματα, τέσσερις δηλώσεις. τέσσερις αυτές δηλώσεις λέγουν ότι η γεωγραφία καταρχάς της Ένωσης αλλάζει. Δεύτερον, οι κοινωνικές διαφοροποιήσεις δυστυχώς και ανισότητες εξακολουθούν να υπάρχουν. Και τέλος η πολιτική παρόλα αυτά δουλεύει. Να ξεκινήσω με την πρώτη διαπίστωση ότι αλλάζει η γεωγραφία της Ένωσης. Αυτό το οποίο δείχνει η έκθεση είναι ότι υπάρχει σύγκληση. Τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες ε, πράγματι εξελίσσονται, αναπτύσσονται. Υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα φυσικά για να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχουν διαφοροποιήσεις, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της Ευρωζώνης και βλέπετε σε ορισμένες ε, περιοχές της Νότιας Ευρώπης και όχι μόνο της Νότιας υπάρχουν δυσκολίες οι δυσκολίες αυτές ε, οφείλονται στο επίπεδο βιομηχανικής εξειδίκευσης, στο επίπεδο κατάρτισης του εργατικού δυναμικού, στη συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας σε παρακμάζοντες τομείς, είναι η λεγόμενη παγίδα του ενδιαμέσου εισοδήματος Νομίζω ότι οι περιοχές αυτές δεν είναι ούτε ικανές να ανταγωνιστούν με τις υπόλοιπες, διότι δεν έχουν την καινοτομική δυνατότητα να το κάνουν και δεν μπορούν φυσικά να ανταγωνιστούν και με τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, διότι έχουν υψηλότερο κόστος εργασίας. Συνεπώς Αυτά λέγει η έκθεση και νομίζω ότι το πιο σαφές μήνυμα είναι ότι αλλάζει η γεωγραφία της Ένωσης και ως εκ τούτου και οι πολιτικές θα πρέπει να εξελιχθούν έτσι ώστε να αντικατοπτρίσουν τη διαδικασία αυτή. Η δεύτερη διαπίστωση είναι ότι παραμένουν και εμένουν οι κοινωνικές ανισότητες. Η απασχόληση φυσικά αυξάνεται, η ανεργία μειώνεται, όλα αυτά είναι αλήθεια αλλά αυτό δεν κρύβει το τι συμβαίνει δηλαδή ακριβώς όταν κάνει κάποιος κάνει ένα μικρό zoom βλέπει ότι υπάρχουν κάποια θέματα στον τομέα των κοινωνικών ανισοτήτων ε, σε ορισμένους τομείς η ανεργία είναι εξίσου υψηλή όπως και πριν από την αρχή της κρίσης και η κοινή αποδοχή των μέτρων για την απασχόληση είναι πάρα πολύ χαμηλή. Το τρίτο, η τρίτη παρατήρηση είναι ότι τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλο και περισσότερο γίνεται ευαίσθητη στο ότι απαιτείται ισχυρή διαχειριστική δυνατότητα και ικανότητα. Γι' αυτό δημιουργήσαμε και τις υπηρεσίες υποστήριξης προς τις περιφέρειες κυρίως Γι' αυτό ακριβώς έχουμε διαπραγματευτεί με ορισμένα κράτη-μέλη κάποια σχέδια για αδικητικού τύπου μεταρρυθμίσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνεται όλο και περισσότερο. Ε, βλέπετε στην έκθεση τη σύνδεση της διοικητικής επίδοσης με, τις ε, λεγόμενες, ε, με τους λεγόμενους δείκτες αποτελεσματικότητας του θεσμικού τομέα. Και η τελευταία διαπίστωση είναι ότι η πολιτική μας είναι αποτελεσματική, δουλεύει. Αρκετά, ε, αρκετά σχεδιαγράμματα δείχνουν ότι έχουν υπάρξει σαφείς βελτιώσεις σε πολλά Είναι η μοναδική πολιτική η οποία διατηρεί σε ανεκτό επίπεδο την δημόσια επένδυση στα κράτη-μέλη κατά τη διάρκεια των προηγούμενων χρόνων, των χρόνων της κρίσης. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ρόλος τον οποίο έπαιξε η πολιτική αυτή ήταν καθοριστικός, αλλά και η αποτελεσματικότητα της πολιτικής αυτής είναι κάνουν, εξαρτάται από το τι κάνουν και οι τοπικές κυβερνήσεις και αν ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση. Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω μία απλή δήλωση. Τελικά, η ουσία είναι ότι θα πρέπει να είμαστε ικανοί να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, η λεγόμενη γεωγραφία της δυσαρέσκειας, τι έχει συμβεί και τι θα συμβεί και πέραν του εθνικού επίπεδου, ακόμα και πέραν του περιφερειακού επίπεδου, ε, γιατί υπάρχουν ανισότητες και στο εσωτερικό των ε, περιφερειών, στο εσωτερικό των αστικών συγκεντρώσεων, στο εσωτερικό των αγροτικών περιοχών και της υπαίθρου. Υπάρχουν ε, θύλακοι στέρησης, υπάρχουν θύλακοι κοινωνικού αποκλεισμού. Συνεπώς λοιπόν αυτά είναι θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν στα πλαίσια της εδαφικής διάστασης των τάσεων των οικονομικών και αν θέλουμε πράγματι να εφαρμόσουμε σωστά τις πολιτικές μας, έχουμε σε αυτά τα οποία έλεγε ο Επίτροπος Έτιγκερ, να υπάρξει δηλαδή μια σωστή ευρωπαϊκή πολιτική για να ανταποκριθεί στα θέματα αυτά. Ευχαριστούμε. Κύριε Μόνφορ, θέλετε το λόγο. Όχι. Σκιώδης εισηγητές. Κύριε Αμπρέσο, πρώτη. Eh, eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζουλό και τον δόκτωρ Ντεμικέλης. για τα όσα μας είπαν ε, όσον αφορά τον εισηγητή και για τα όσα έκανε ο κύριος Δεμικέλης, ε, ο δόκτωρ Δεμικέλης. Ε, πράγματι αυτή η νέα πολιτική συνοχή, η μελλοντική πολιτική συνοχής ε, θα είναι η πρώτη μετά από μια δεκαετία βαθύτατης κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάλυση λοιπόν των όσων συνέβησαν σε αυτό το διάστημα θα είναι πιστεύω πολύ σημαντική ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά τον μελλοντικό προγραμματισμό. Εδώ δεν θα πρόκειται πλέον μόνο για πολιτική σύγκληση μεταξύ ε, περισσότερο και λιγότερο εξελιγμένων περιφερειών. Θα είναι μια πολιτική η οποία θα εξετάζει σε βάθος τι συνέβη κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Κρίση η οποία ξεκίνησε από τον οικονομικό τομέα με τρόπο που κατέστρεψε μια οικονομία που υπήρχε στο παρελθόν, που στην Ευρώπη είχε υπάρξει πλέον απερχαιωμένη σε σχέση με άλλες πιο ανταγωνιστικές οικονομίες ε, και την οποία ε, τροποποίησε και άλλαξε, μετέβαλε τελείως η κρίση. Η νέα γεωγραφία λοιπόν της Ευρώπης δεν μπορεί λοιπόν ε, κατά κανένα τρόπο να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στο εισόδημα και στα έσοδα. Θα πρέπει, όπως λέει η έκθεση, αλλά ίσως η, περιλήψη της έκθεσης να μην είναι τόσο ευνόητη. Ε, πρέπει να μπούμε σε βάθος ε, στην κατάσταση που έχει η Ευρώπη για να καταλάβουμε ποιες τάσεις υπάρχουν οι οποίες οδηγούν σε μεταβολές, σε ανάπτυξη ή σε ε, οπισθοχώρηση ή σε προβλήματα γιατί για τον επερχόμενο προγραμματισμό για να γίνει σωστά πρέπει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε μετά από μια δεκαετία σοβαρότερης κρίσης, κρίσης άνευ προηγουμένου για την μεταπολεμική Ευρώπη. Κανείς δεν θα είχε ποτέ φανταστεί ότι θα περνάγαμε θα περνάγαμε μια δεκαετία σχεδόν ε, υποπληθωρισμού με αποτελέσματα τραγικά για πολλούς τομείς. Αυτό που προκύπτει λοιπόν, ε, και εγώ τώρα αυτά που τα λέω τα βασίζω στην πρώτη μου ανάγνωση, θα συζητήσουμε όμως και με τον εισηγητή, ε, με την έκθεσή του. Πιστεύω λοιπόν και εγώ ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ε, στις πλέον ανεπτυγμένες περιοχές της Ευρώπης που είναι όμως πιο αδύναμες ανταγωνιστικά. Τι συνέβη, διότι ε, σε αυτή τη δεκαετία της λιτότητας, ε, σε συνδυασμό με την κρίση, σε πολλές χώρες μειώθηκαν οι επενδύσεις και συνεπώς ε, οι δυνατότητες καινοτομία έρευνας. Σημαντικές λοιπόν περιοχές της Ευρώπης με μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες, ανέκαθεν εύπορες, κατέστησαν, εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους που υπάρχουν, ε, αδύναμες. Και αυτό τροφοδοτεί τη θέση που, ε, επί της οποίας συμφωνούμε όλοι ότι η πολιτική πρέπει να αφορά όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Οπότε το θέμα δεν είναι απλά να ανεβάσουμε στο μέσο όρο τους στοχότερους. Το πρόβλημα είναι ότι στο μέσο όρο βρίσκουμε ξαφνικά μια κρίση, πολλές κρίσεις σοβαρές που αν δεν τις προσέξουμε, αν δεν μεριμνήσουμε για αυτές, θα ε, οδηγήσουν σε ε, οπισθοχώρηση. Μετά τώρα υπήρχε το ζήτημα του ότι και εντός των ε, εύπορων περιφερειών εμφανίζονται φαινόμενα πόλωσης. Και όταν λέω πόλωση, δεν είμαι απόλυτα ακριβής, γιατί έχουμε το πρόβλημα των αγροτικών περιοχών, ε, ορεινών ε, και τα λοιπά, που έχουν ε, πολλά χαρακτηριστικά διαφορετικά, όπου η κρίση των δημόσιων οικονομικών και οι περικοπές και άλλοι λόγοι, πολύ περίπλοκοι, οδήγησαν και οδηγούν σε απερίμωση των υπηρεσιών Οπότε στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας μην ξεχνάμε ότι ε, η ύπεθρος, ε, τα βορεινά, οι βορεινές περιοχές είναι πάνω από το 70% της επικράτειάς μας. Οπότε μιλάμε για περίμωση, για ερήμωση. Εντός των πόλων αντιθέτως, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι πόλος το φαινόμενο, εντός των πόλων λοιπόν ε, παρατηρούμε ένα σημαντικότατο πρόβλημα περιφερειών και εδώ υπάρχουν δομικοί λόγοι. Η Ευρώπη ανοικοδομήθηκε πολύ γρήγορα, ολόκληρη στη μεταπολεμική εποχή. Αφού είχαν καταστραφεί οι πόλεις ε, κατά τον πόλεμο, ανοικοδομήθηκε μετά τον πόλεμο, μετά τον πόλεμο. Και τώρα έχουν περάσει πλέον 70 χρόνια από τον πόλεμο. Και είναι σαφές ότι αυτές οι ζώνες που ανοικοδομήθηκαν γρήγορα επειδή υπήρχε αυτή η απέτηση να δοθούν κατοικίες ε, στον κόσμο έχουν ε, παλιώσει, έχουν αποδυναμωθεί, δε, τους λείπουν ε, βασικές υπηρεσίες ε, και απαιτούν τεράστιες επενδύσεις. Αυτά είναι τα άλλα ζητήματα ε, που θεωρώ σημαντικά. Πιστεύω ότι εμείς, παρότι το χρονοδιάγραμμα, όπως είπε ο εισηγητής, είναι πολύ δύσκολο και περιορισμένο, θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε προσοχή σε αυτά τα ζητήματα, διότι από τη μία πλευρά χρειάζονται πόροι, από την άλλη όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά και αυτές τις διαφορές. Θα μπορούσαμε ενδεχομένω ε, να καταστήσουμε πιο ευέλικτη και πιο προσαρμόσιμη ε, την πολιτική συνοχή για τι περιφέρειες. Να μην λέμε ότι η ψηφιοποίηση χρησιμεύει για όλου. Το πρόβλημα είναι ότι η ψηφιοποίηση δεν πραγματοποιείται και δεν υλοποιείται με τον ίδιο τρόπο στις πόλεις και στην Ήπεθρο. Και αυτό ισχύει και για άλλε πολιτικέ, πολλέ μάλιστα. Η ψηφιοποίηση δεν είναι ένα παράδειγμα, οπότε χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία ε, στον τρόπο, στι προποθέσει ε, εφαρμογής ε, των ε, στόχων. Πραγματικά υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τις δυνατότητες ε, παρέμβασης των ε, περιφερειακών και τοπικών φορέων. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν αρκεί να προσφέρουμε απλά κάποιο είδος ε, τεχνικής υποστήριξης. Χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε ριζικά εντός των κρατών το εξής πρόβλημα του πώς οι περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις θα καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις μέσω συνεργασίας, ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές ενδεχομένως, ανταλλάσσοντας εμπειρογνώμονες γνώσεις, αλλά και προσφέροντας κατάρτιση, πιο ε, απτή στήριξη ε, που να καλύπτει τις απαιτήσει τους και τις ανάγκες τους. Το τελευταίο που ήθελα να πω αφορά την ενεργεία η ενεργεία σχετίζεται κατά μία έννοια με την κρίση, με τη μείωση του εισοδήματος που θα ε, βελτιωθεί με την έξοδο από την κρίση αλλά που και διαρθρωτικά προβλήματα. Από τη μια πλευρά η αβεβαιότητα της εργασίας ε, στη Γερμανία αυτό δημιουργεί, ε, στη εντάσεις η συζήτηση σήμερα ε, είναι ότι πολλές από τις νέες δουλειές που δημιουργούνται είναι αβέβαιου τύπου. Ε, είναι δουλειές low cost, χαμηλού κόστους. Σήμερα ε, αυτή η τάση low cost, χαμηλού κόστους, φαίνεται να είναι κανόνας και στην εργασία. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα διερμηνίας? Ναι, όχι, εντάξει. Δεν έχουμε πρόβλημα με την διερμηνία. Με το χρόνο έχουμε πρόβλημα, λέει ο πρόεδρος. Αυτά ναι, τελειώνω σιγά σιγά, λέει η κυρία Μπρέσο. Λοιπόν, όπω είπα, αυτές οι εργασίε χαμηλού επίπεδου και η χαμηλή ε, υποστήριξη που προσφέρεται γενικά ε, σε πολλούς ε, τομείς, μάλιστα το δούμε να συνεχίζεται αυτό. Για να καινοτομήσουμε και να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί υπάρχει κίνδυνος να μειωθούν ακόμη περισσότερο τα επίπεδα απασχόλησης. Οπότε δημιουργείται το πρόβλημα ε, δημιουργίας θέσεων εργασίας που δεν σχετίζονται, σχετίζονται μόνο με την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και σε εποχές όπου κινούμαστε προς την αυτοματοποίηση, τη χρήση περισσότερων ρομποτικών μηχανισμών, ε, τίθεται το θέμα του πώς θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και θα δοθούν τα μέσα διαβίωσης στους ανθρώπους. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Επόμενος κοιόδης ε, είναι η κυρία Τόμασιτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερος που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της έλλειψης εμπιστοσύνης. Υπάρχει ένα πρόβλημα έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ δηλαδή εθνικών και περιφερειακών αρχών. Υπάρχει ένα πρόβλημα λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι καλό που έχουμε αυτή την πολιτική γιατί βρισκόμαστε σε εποχή παγκοσμιοποίησης και δεν πρέπει κανείς να μείνει πίσω υπάρχουν ε, κάποιες περιφέρειες που αναπτύσσονται, άλλες όχι. Υπάρχουν πολλές περιφέρειες που προσέγγισαν το Μεσόρο, αλλά έπεσαν σε παγίδα τελικά, γιατί οι δημόσιες επενδύσεις στην Ένωση είναι μικρότερες σε σχέση με πριν την κρίση. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να αναφερθεί στην έκθεση. που μελετά τι μελλοντικέ προοπτικέ. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη επίση οι κλιματικέ αλλαγές, η ψηφιακή μετάβαση και η σύγκληση των περιφερειών. Περιφέρειες που συχνά έχουν να αντιμετωπίσουν ε, απόλυτε θέσεις εργασίας, θέσεων εργασίας, κλείσιμο βιομηχανιών κτλ. κτλ. Πρέπει να στηρίξουμε τις περιφέρειες αυτές για να μπορέσουν να επιβιώσουν στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Πρέπει να του βοηθήσουμε να δημιουργήσουν θέσει εργασία και ανάπτυξη. Ορισμένε περιφέρειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παραδείγματα επιτυχημένα και αποδεικνύουν ότι πρέπει να επενδύσουμε στην καινοτομία και στην ψηφιοποίηση. Βεβαίως, επιχειρήσεις και τα κέντρα καινοτομίας ε, και έρευνα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ του. Στην παραδείγματο χάρη, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη μαζική φυγή. Έξοδο, μαζική έξοδο. Και βέβαια μεγάλο πρόβλημα μεταναστευτικό. Έχουμε πολύ ψηλή ανεργία μεταξύ των νέων επίσης. Μια άλλη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι οι διαθετικές μεταρρυθμίσεις σε πολλά κράτη-μέλη. Βελτίωση δημόσιας διοίκηση είναι ένα άλλο θέμα. Βελτίωση του ανταγωνισμού και της ανταγωνιστικότητας. Στην 7η έκθεση συνοχή, λοιπόν, πρέπει νομίζω να δείξουμε καλύτερα τη σχέση που έχουν ρυθμίσεις οικονομική πολιτική και η στήριξη δημοσιονομική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή έκθεση και δίδεται προσοχή στην ανάπτυξη των περιφερειών, ιδιαίτερα στις μεθοριακές περιοχές. Το θέμα της ανεργίας είναι πάντα πιο υψηλό από ε, πριν από την κρίση. Απαιτούνται μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας έτσι ώστε να ανεπτυχθούν και οι δυνατότητες της διαμεθοριακής απασχόλησης. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα ήθελα να δω στην έκθεση Ζουλό είναι σαφές ότι δεν επενδύουμε επαρκώς στον τομέα της καινοτομίας, απόκτησης ικανοτήτων, ψηφιακών ικανοτήτων, υποδομών, ενεργειακής αποδοτικότητας, ανανεώσιμων και ε, καθαρών μεταφορών. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε, θα αντιμετωπίσουμε το θέμα των ε, εκπομπών ιδιαίτερα για την πολιτική μας μετά το 2020 υπάρχουν πολλές απορίες, δεν μπορούμε να τα κάνουμε για μια όλα και πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας. Επίσης πρέπει και η διακυβέρνηση να βελτιωθεί. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να επενδύσουμε σε διαφορετικές μεταρρυθμίσεις εφόσον πράγματι θέλουμε να προχωρήσουμε. σε μια σελίδα της έκθεσης υπάρχει ένας πίνακας που δείχνει την αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης και βλέπει κανείς το 90, 90, η διαφορά από το 96 μέχρι το 2015 σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία είναι πάντα τελευταίες. Θα πρέπει να το συνδέσουμε αυτό με όλες τις εμπειρίες τις οποίες είχαμε μέχρι τώρα από τις επισκέψεις μας στη Σοφία και στο κλούς και να δούμε ακριβώς το τι συμβαίνει. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με μια πολιτική συνοχή επενδύοντας σε χώρες όπως η Βουλγαρία με τα ίδια ακριβώς χρήματα όπου οι συστάσεις αναχώρα δείχνουν ότι υπάρχει έλλειψη στην δυνατότητα συλλογής φόρων σαν παράδειγμα σε κάποιες χώρες. Ε, δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση αυτή, πρέπει να διορθωθεί. Πρώτα λοιπόν διαφθρωτικές μεταρρυθμίσεις, μετά βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης μέσω της εφαρμογής των ειδικών συστάσεων, γιατί δεν μπορεί από τη μία να μην μπορείς να συλλέξεις τους φόρους και από την άλλη να ζητάς χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο δεν θα κατανοήσει ο Ολλανδός φορολογούμενος. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος των Πρασίνων. Ρόπε. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Η έκθεση η φετινή είναι ένα πολύ καλό έγγραφο αλλά περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία τα οποία είναι ανησυχητικά. Από τη μία πλευρά είναι θετικό το ότι μειώνονται οι διαφορές μεταξύ των διαφορών περιφερειών, ότι βελτιώνεται το επίπεδο των φτωχότερων και ότι διαπιστώνεται κάποια οικονομική ανάπτυξη. Αλλά αν δούμε τα στατιστικά στοιχεία για την περίοδο 2000 έως 2015, το ΕΠ των λιγότερων ανεπτυγμένων περιοχών πλησίασε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι αναπτύχθηκε, αυξήθηκε η παραγωγικότητα αλλά οι θέσεις απασχόλησης μειώθηκαν σε αυτές τις περιοχές. Πρέπει να πούμε πίσω ότι σε πολλές από αυτές τις περιοχές το κατακεφαλήν ΑΕΠ δεν φτάνει στο επίπεδο πριν την κρίση. Επίσης είναι ανησυχητικό το ότι οι πολίτες μας αξιολογούν ε, την πολιτική συνοχή όχι πάντα θετικά. Κατά την άποψή μου, η επιτυχία της πολιτικής συνοχής ε, μπορεί να μετρηθεί από το πόσο επιθυμούν οι πολίτες να παραμείνουν στις περιοχές τους. Αλλά ε, κοιτώντας τα δεδομένα παρατηρούμε ότι σε πολλές περιφέρειες όπως λέμε στα λιθουανικά, οι πολίτες παίρνουν τα πόδια τους και φεύγουν. Φεύγουν τρέχοντας από αυτές τις περιοχές. Πρέπει να βρούμε για ποιο λόγο φεύγουν οι πολίτες από τις περιοχές αυτές. Και να βρούμε έναν τρόπο να μειώσουμε αυτές τις αναχωρήσεις. Αυτό θα μας επιτρέψει να αξιολογήσουμε την επιτυχία ή αποτυχία της πολιτικής συνοχής. Θα ήθελα λοιπόν να, ο, ο εισηγητή να επικεντρωθεί περισσότερο στην εξέβριση αυτών των αιτιών και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω ε, για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μανταμάτο, έχω ε, κάποιες σκέψεις για αυτή την έβδομη έκθεση, η οποία πιστεύω έχει σημαντικές αντιφάσεις. Απ' τη μια αναγνωρίζει ότι η πολιτική συνοχή είναι η βασική επενδυτική πολιτική της Ένωσης, με επενδύσεις 8,5% ε, που ανεβαίνει στο 50% για κάποιες άλλες χώρες. Όπως ξέρουμε αυτές οι επενδύσεις συμβάλλουν για ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά. Από την άλλη όμως και αναγνωρίζοντας ότι οι συνολικές επενδύσεις ε, ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν μειωθεί κατά την κρίση και δεν έχουν αυξηθεί σχεδόν καθόλου από τότε, δεν καταλαβαίνω πώς διαπιστώνεται στην 7η έκθεση συνοχής. Δεν λέγεται τίποτα για το άρθρο 23 και για τη σχέση μεταξύ πολιτικής συνοχής ε, και εκτός Ευρώπης. Καμία πρόταση αλλαγής λοιπόν. Πώς είναι δυνατόν όλο αυτό. Παρότι είδαμε ένα σωρό πράγματα με την Ισπανία και την Πορτογαλία πέρυσι, τίποτα, καμία κύρωση δεν επιβλήθηκε. Έχουμε ακόμα χρόνο και ελπίζω να το κάνουμε κατά τι διαπραγματεύσει, να εκφράσουμε μια ισχυρή θέση ω συνομοθέτε. Πριν από ένα μήνα στο Ευρωκοινοβούλιο στην Ολομέλεια, η πλειοψηφία εκφράστηκε κατά τη οικονομική, ερεσιμότητα, ε, μακροοικονομικής Έτσι πρέπει να δράσουμε. Δεν καταλαβαίνω πως η Κομισιόν δεν έλαβε υπόψη τη θέση μας. Εγώ για χιλιοστή φορά θέλω να καλέσω τους συναδελφούς να δουν το πρόβλημα στη ρίζα του, να καταλάβουν πώς συνδέεται το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και η πολιτική συνοχής και να καταργηθούν όλες οι κυρώσεις που είναι πολύ τιμωρητικέ και περιτές για τις ε, περιφερειακές και τοπικές ε, αρχές. Η πολιτική συνοχή δεν είναι αυτή που δημιουργεί το χρέος. Αν ξεκινήσουμε όμως από επεκτατική επενδυτική πολιτική θα μπορούσε να αποτελέσει τη λύση. Πολλά θέματα πρέπει να αναλύσουμε και να σκεφτούμε όταν θα έχουμε το σχέδιο εκτίση του συναδέλφου, ούτω θα πράξουμε κυρίω όσον αφορά την ανεργία των νέων και την απερίμωση ορισμένων περιοχών. Για να κλείσω αυτή η πρώτη ανταλλαγή, πιστεύω πρέπει να μας θυμίσει ότι τόσο το έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών, όσο και η παρούσα έκθεση για το ζήτημα αυτό, υποστηρίζουν και τα δύο ότι η χαμηλή θεσμική ποιότητα ε, θέτει σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα, της επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη. Και τα δύο έγγραφα δίνουν έμφαση στη βελτίωση της διακυβέρνησης, ε, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στην ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων. Εγώ λοιπόν συμφωνώ με τα μέτρα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δημοσίων διοικήσεων, της, ικανότητές τους, να βοηθήσουν του πολίτες. Οι μεταρρυθμίσεις λοιπόν πρέπει να γίνουν για να βελτιώσουν τα μέτρα και από δημοσιονομική άποψη. Αλλά προσοχή, μην προσθέσουμε επιπλέον αιρεσιμότητες που θα ε, τιμωρήσουν τους δικαιούχους. Ε, οι ιδιωτικοποίησεις διαρθρωτικές όπως έγιναν σε πολλές χώρες όπως και στη δική μου στους τομείς της εργασίας, της εκπαίδευσης δεν δημιουργούν μόνο ε, προβλήματα στην κοινωνική συνοχή αλλά δημιουργούν και προβλήματα αύξησης των χασμάτων σε οικονομικό, εδαφικό και κοινωνικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εμείς. Δεν έχω κάποιον άλλο σε κατάλογο των ομιλητών. Α, έχω. Συγγνώμη, τον κύριο Νοβάκοφ έχω. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχά θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ζούλο για τη σκληρή του δουλειά και την αφοσίωσή του. Είμαι βέβαιος ότι το αποτέλεσμα θα είναι όπως πάντα καλό. Δεν μπορώ να πω ότι η 7η έκθεση συνοχής πηγαίνει πολύ ξεκάθαρα προς ε, μια κατεύθυνση, είναι αντιφατική σε κάποια σημεία. Ενώ σε κάποια άλλα δίνει συγκεκριμένες προτάσεις. Εγώ θα ήθελα να είναι πιο πολλές σε συγκεκριμένες προτάσεις. Ελπίζω να συμβεί αυτό στην 8η έκθεση συνοχής. Σε ό,τι αφορά το μέλλον της πολιτικής συνοχής, πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές το έβδομο πλαίσιο συνεχής μπορεί να είναι ίσως η βάση, δηλαδή να αντλήσουμε διδάγματα για το μέλλον. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει με το επίπεδο ΝΑΤΣ 3, μήπως πρέπει να επιλέξουμε άλλα κριτήρια για τις επιλέξιμες περιφέρειες, τι θα γίνει με τις συστικές στάσεις αναχώρα κτλ. κτλ. Όταν όμως αρχίζουμε συγκεκριμένα να βλέπουμε τα παραδείγματα πρέπει να έχουν υπόψη μα ότι δεν δίνουν την πλήρη εικόνα. Αναφέρθηκε μια τη χώρα που γνωρίζω πολύ καλά. Ότι δεν υπάρχουν αρκετά φορολογικά έσοδα. Διπλασιάστηκε το ΑΕΠ από τότε που γεννάμε μέλο τη Ένωση. Άρα εγώ νομίζω ότι τα πάμε καλά. Επίσης, είχαμε και πλεόνασμα στο προορισμό πρόσφατα. Λόγω και βελτίωση τη ύπραξη φόρων. και σε επισκέψεις στη Βουλγαρία οι προσωπίες έχουν διαπιστώσει πολλάκις ότι χρησιμοποιεί επαρκώς η χώρα τα κονδύλια και υπάρχουν απτά αποτελέσματα. Και οι συστάσεις αναχώρα λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη στην Βουλγαρία. Αυτό και δεν είχαμε ποτέ δημοσιονομικό έλλειμμα 3%. Δεν θέλω να αναφέρω κάποια συγκεκριμένη κυβέρνηση, αλλά εμείς ακολουθούμε τους κανόνες του να μην υπερβούμε το 3%. Άλλες όχι. Γιατί η έκθεση πάντως είναι καλή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση. Δεν είναι και βίβλος όμως. Άρα πρέπει να βλέπουμε την γενικότερη εικόνα όταν καταλήγουμε στα συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Κύριος Χάουαρντ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. η πολιτική συνοχή όσο υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τι μεγαλύτερε επιτυχίε τη Ευρώπη. Και αυτό δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Παρά τις δυσκολίες, βράχει πρόθεσμα. Αλλά αυτό δημιουργεί και μεγαλύτερε προσδοκίε για το πώ θα συνεχίσει να αποδίδει αποτελέσματα η πολιτική αυτή και στο μέλλον. Χαιρετίζω την έκθεση και τα σχόλια ε, τη Κομισιόν και του Επιτρόπου έτοιμη συγκεκριμένο, ο οποίο είπε κάτι πολύ σημαντικό μεταξύ άλλων. Δηλαδή, οι πλούσιε περιοχέ Ένωση. Πόσο ασχολούνται ή δεν ασχολούνται με την πολιτική συνοχή και πόσο συνεισφέρουν. Σε δύο επίπεδα. Πρώτον, τι γίνεται με τι πλούσιες περιφέρειες. Είναι δύσκολο να κάνει φτωχό σε μια πλούσια περιφέρεια. Υπάρχουν φυλάκε φτώχεια και κοινωνική εξαθλίωση σε όλε τι πλούσιε περιφέρειε. Πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι περιφερειακέ κυβερνήσει πρέπει να επιμείνουν και πρέπει να τις έχουμε υπόψη αυτές τις περιοχές. Αλλά και οι ίδιες περιφέρειες πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο γιατί ανταγωνίζονται σε διεθνέ επίπεδο και θα πρέπει να αναπτύξουν τις εμπορικέ δραστηριότητες, οι λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και γενικώ να υπάρχει καλύτερη εμπορική σχέση μεταξύ φτωχότερων και πλεισότερων περιφερειών. Αυτό απαιτεί και μια πιο ευφύ προσέγγιση στην πολιτική υποδομών που πολλές φορές ε, είναι μοχλός συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ψηφιακέ υποδομές πρέπει να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο από ότι οι υλικές υποδομές κατά το παρελθόν, διότι αυτός είναι ο δρόμος του μέλλοντος. Τρίτον, η αύξηση της δυνατότητας απορρόφησης των πολιτικών όπως πολιτική απασχόληση λοιπά. Είναι κάτι που το ακούω συνεχώς εδώ από τις αρχές που επιζητούν συμμετοχή στα προγράμματα της Ένωσης. Να είναι πιο εύκολο αυτό, λιγότερο γραφειοκρατικό. Αλλά βέβαια ταυτόχρονα να υπάρχουν τα εχέγγυα και ασφαλιστικές δικλείδες. Αυτή είναι μεγάλη πρόκληση για την αντιμετώπιση της ανεργίας για παράδειγμα. Επίσης η Επιτροπή προϋπολογισμών ναι, μέχρι τις 4 το πρωί το Σαββάτ με τον Επιτρόπο Έντιγκερ κατάφεραν τελικά να βρουν ένα συμβιβασμό. Και σίγουρα θα είναι δύσκολα τα νούμερα. Η ευφύς χρηματοδότηση θα ενταχθεί. Και ίσως τελειώσω με κάτι απεσιόδοξο, αλλά κάτι που πρέπει να το πω παρόλα αυτά με την ε, φορολόγηση και τους πόρους ε, δεν νομίζω ότι θα έχουμε επαρκή πολιτική συνεχίση. Είναι αυταπάτη. πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα χρηματοδοτικά μέσα και όχι να δίνουμε επιδοτήσεις και ενισχύσεις. Πρέπει να γίνει σοβαρή σκέψη επ' αυτών. Αλλά γενικώ νομίζω ότι η πολιτική συνοχή είναι από τι πιο επιτυχημένε πολιτικέ και ελπίζω να συνεχίσει να είναι. Ευχαριστώ κύριε Βανίστελ Θέλετε το λόγο. Θα είμαι σύντομο. Μια και συζητήσαμε με τον Επίτροπο για τον προπολογισμό. θα προσπαθήσουμε την έκθεση αυτή την πολύ πλούσια ιδιαίτερα στον τομέα της εδαφικής συνεργασίας σε διαμεθοριακές περιοχές. Υπάρχουν πολλά τα οποία έχουμε να δούμε. Η έβδομη λοιπόν έκθεση σύνοχης ίσως να αποτελέσει την επόμενη φάση του κανονισμού για τον κανονισμό. Είχαμε έτσι και αλλιώς τα θεμέλια με την έκθεση της κυρίας Βέστφαλ και μπορούμε ακριβώς να δούμε τι λέει το 7ο πρόγραμμα, η 7η έκθεση, ε, για να γίνουμε πιο επακριβείς. Ο κίνδυνος είναι να ξεκινήσουμε με πάρα πολλές τροπολογίες, να οδηγήσουμε τα πράγματα από την αρχή, για μια ακόμη φορά. Να ξεκινήσουμε από το μηδέν, όπως παλαιότερα που ήμουν εγώ εισηγητής. και αναφερθήκαμε στις εταιρικέ συμφωνίες ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη ή καλύτερα τις περιφέρειες. Και μετά περάσαμε στα θεμέλια και μετά περάσαμε στην απλούστευση. Το μεγαλύτερο λάθος λοιπόν είναι να διπλασιάζουμε και να τριπλασιάζουμε τα πάντα. Ίσως μπορούμε να το συζητήσουμε το θέμα και στους συντονιστές δεν θα πρέπει να φεύγουμε προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά θα πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τα μηνύματα που μας έδωσε ο Έτιγκερ σήμερα το πρωί. Υπάρχει μια ευκαιρία και υπάρχει μια μεγάλη έκθεση η οποία μπορεί να μας απασχολήσει και είναι αυτή. Είναι κάτι το οποίο πράγματι εντάσσεται στο χρονοδιάγραμμα που έχουμε μπροστά μας έτσι ώστε να μπούμε στη νέα περίοδο, μέχρι το τέλος δηλαδή της περίοδου αυτής, we should not deep our our our debates deeper and deeper and deeper. Και θα πρέπει να εμβαθύνουμε λοιπόν στα θέματα που μας ενδιαφέρουν για να επιβάλλουμε την πολιτική συνοχή σε ένα ευρύτερο επίπεδο και να φτάσουμε στην Ολομέλεια. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα κάνουμε τις πολιτικές μας επιλογές σε σχέση με την έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θα ήθελα το λόγο. Ο κύριος Μονφόρ και ο κύριος Ντεμικέλης θα ήθελαν πάλι να πάρουν το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο πάρα πολύ σύντομες παρατηρήσεις. Η πρώτη. Συζήτηση για τις διαφορετικές αλλαγές, αλλαγές γενικότερα, μεταρρυθμίσεις γενικότερα. Έχω την αίσθηση ότι η εποχή κατά κάποια μια περίοδο που η περιφερειακή πολιτική ε, ήταν ανεξάρτητη ουσιαστικά από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έχει περάσει πια. Όταν μιλάμε για μεταρρυθμίσεις το θέμα είναι να δούμε τι είδους μεταρρυθμίσεις συζητάμε. Και εδώ υπάρχουν πράγματα που μένει να γίνουν. Σαν παράδειγμα διοικητική ικανότητα, θεσμικά όργανα. Μιλάμε για μεταρρυθμίσεις τις οποίες ήδη έχουμε σιγά σιγά περάσει με την εκ των προτέρων ερεσιμότητα που ήταν απαραίτητες για να δείξουμε στους επενδυτές ότι είμαστε σοβαροί. Ή μιλάμε για ευρύτερες μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν άμεση σχέση με την πολιτική συνοχής και για τις οποίες θα υπάρχει ανάγκη για μια συζήτηση έτσι ώστε η πολιτική αυτή να μην μετατραπεί σαν ένα επιπλέον δημοσιονομικό μέσο επιβολής κυρώσεων στα κράτη-μέλη τα οποία δεν αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρα στις υποχρεώσεις τους. Νομίζω λοιπόν ότι, και έρχομαι στο δεύτερο σημείο, ότι στα πλαίσια της συζήτησης για το δημοσιονομικό κομμάτι του νέου ε, πλαισίου Υπάρχει μια περίεργη διχοτομία ανάμεσα στις επενδύσεις από τη μία και τη συνοχή από την άλλη. Γιατί συμβαίνει αυτό, η, συνοχή είναι οι επενδύσεις. Δεν είναι κάτι το ξεχωριστό σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει η Ένωση στον τομέα των μεταρρυθμίσεων, της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, της καταπολέμησης των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος. Και αυτό το οποίο πρέπει να δείξουμε είναι ότι η πολιτική αυτή έχει μια διαφορετική διακυβέρνηση αν θέλετε και η γεωγραφία της ε, ε, είναι κάπως διαφορετική από τα άλλα μέσα, αλλά κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Αντιμετωπίζει ακριβώς τις ίδιες προωθεί, μάλλον τις ίδιες προτεραιότητες. Αυτό θα πρέπει λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε και να μην δίνουμε την εντύπωση ότι η πολιτική συνοχή είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό από τις συζητήσεις έχουμε, που έχουμε κάνει μέχρι τώρα σχετικά με τις προτεραιότητες. Και τώρα το χρονοδιάγραμμα. Είναι σαφές ότι ό,τι μπορεί να κάνει κανείς για να επιταχύνει τα προγράμματα αυτά είναι σωστό. Η περίοδος επιρροής είναι τώρα και για τους επόμενους δύο-τρεις μήνες. Πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατασταλάξει στις τελικές της προτάσεις, δηλαδή τον μήνα Μάιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζουό. Έχετε το λόγο κύριε Ζουλό. Σύντομα πρόεδρε. Να ευχαριστήσω ξεκινώντας τους εισηγητές, τους κοιόδους που πήραν το λόγο και όλους τους συναδέλφους που εξέφρασαν τις προτεραιότητές τους, τις ιδέες τους και τις ε, απόψεις τους γενικότερα να ευχαριστήσω και τον κύριο Ντεμικέλης και για το τελευταίο σημείο που τέθηκε το θέμα του χρονοδιαγράμματος. Μας υποχρεώνει να πάμε γρήγορα, αλλά συμφωνώ ότι η έκθεση αυτή είναι μια ευκαιρία για να μπορέσουμε να περάσουμε ακριβώς ε, ισχυρά μηνύματα μπαίνοντας ε, και στις γενικές ε, αρχές και στις λεπτομέρειες αυτής της πολιτικής. Εν πάση περιπτώσει εγώ είμαι διατεθειμένος να συνεργαστώ και ε, με τους συνεργάτες μου για να προωθήσουμε τις ιδέες τις οποίες αναφερθήκατε σήμερα. Σας ευχαριστώ. Η βασική ιδέα της ΒΕΤΖ είναι να προετοιμάσει την έκθεση αυτή λοιπόν πριν πάρουμε την πρόταση για το πολιετές δημοσιονομικό, για το νέο πολιετές δημοσιονομικό. Και γι' αυτό ακριβώς εμείς αναφερόμαστε σε ένα χρονοδιάγραμμα του για το Φεβρουάριο ε, του 2018. Οι τροπολογίες ε, θα κατατεθούν στο τέλος Φεβρουαρίου και θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην Ρέτζη τον Απρίλιο. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε την τελική άποψη της Ρέτζη που θα βασίζεται ε, στα συμπεράσματα της 7ης έκθεσης συνοχής διαθέσιμες τον μήνα Απρίλιο. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα προς το παρόν. Ελπίζω ότι ο εισηγητής και οι σκιώδεις θα επενδύσουν ε, σοβαρά στην προσπάθεια για να στηρίξουν την προετοιμασία της έκθεσης αυτής. Σας ευχαριστώ όλους ε, για τη συζήτηση αυτή. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα μας ε, και θα συνεχίσουμε τώρα με την ημερήσια διάταξη. Το επόμενο θέμα είναι τα διάφορα. Υπάρχει ε, κάτι, όχι δεν ε, υπάρχει κάτι. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι η επόμενη συνάντησή μας θα είναι η μέρα 5η 7 Δεκεμβρίου 9 το πρωί και όλη την ημέρα. Λοιπόν, τερματίζεται ε, η συνεδρίαση της, του συνόλου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και να παραμείνουν παρακαλώ στην αίθουσα όσοι συμμετέχουν στη συνάντηση των συντονιστών. Θα συνεχίσουμε με τη συνάντηση των συντονιστών.